Okay, so good morning everybody. Good morning and welcome to the European Parliament. Uh, Καλημέρα και καλώς ήρθατε. Μας συγχωρείτε για τις ε, καθυστερήσεις αυτές λόγω των αυξημένων μέτρων ασφαλείας που αναγκαστήκαμε να λάβουμε στο Κοινοβούλιο λόγω της ε, προβληματικής ε, κατάστασης μετά τις τρομοκρατικές επιθέσεις στο Παρίσι. Γιάννης Ντάνης λέγομαι, είμαι από την υπηρεσία που οργανώνει το σεμινάριο για... Δαρμής. λέγεται ο κύριος, για το άσυλο και τη μετανάστευση. Εδώ πέρα έχουμε την κυρία Ζαβέλα Ταρκάνη, η οποία είναι αρμόδια από την πλευρά του τύπου για την νομοθεσία μετανάστευσης και ασύλου και θα κάνει μια εισαγωγή στο έργο της Επιτροπής ΛΥΜΠΕ των πολιτικών ελευθεριών δηλαδή. Εκ μου Μάρκο Σετερίνο από την εφημερίδα Λαστάμπα, ανταποκριτής από το 2006 με γνώση των ευρωπαϊκών θεμάτων, ο οποίος θα συντονίσει τα πάνελ αργότερα και ο Νταμιάν Καστάνιο βεβαίως ε, επίσης ε, εκ των οργανωτών αυτού του σεμιναρίου. Ξεκινήσαμε χτες, όπως ξέρετε, με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, τον ε, Μάρτιν Σούλτς, και θα συνεχίσουμε σήμερα με ανταλλαγές απόψεων με βουλευτές και μια εκπρόσωπο της ΥΠΑ του ΟΗΕ για τους προσήγες. Επίσης πρέπει να υπογραμμίσουμε πως το σεμινάριο αυτό έχει συγκεντρώσει εδώ 196 δημοσιογράφους ε, από όλες τις χώρες, μεταξύ των οποίων 33 ε, τηλεοπτικούς σταθμούς και 31 ραδιοφωνικούς σταθμούς. Ξέρετε πως ε, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο παίζει σημαντικό ρόλο σχετική νομοθεσία. Αυτή τη στιγμή η αρμόδια οι αρμόδιες ε, επιτροπές εξετάζουν ε, σχέδια νομοθεσίας ε, που αφορούν ζητήματα όπως έναν μόνιμο μηχανισμό ανακατανομής, την χρηματοδότηση και διαχείριση της μεταναστευτικής κρίσης, αλλαγές στο Δουβλίνο, μια κοινή λίστα ασφαλών χωρών προέλευσης, καθώς επίσης τη δραστηριότητα της ε, Frontex και την δημιουργία των ε, hotspots. Πρόκειται για μια εκδήλωση λοιπόν που διοργανώνουμε ε, γι' αυτό όπως και για άλλα σημαντικά ζητήματα. Στόχος είναι να ξεκινήσει μια συζήτηση με εσά και να εξηγήσουμε το τι κάνει το Κοινοβούλιο στο θέμα μετανάστευσης και ασύλου. Ο στόχος μας είναι γενικότερα να ενημερώσουμε τους μουσιογράφους για ζητήματα τα οποία έχουν άμεσο αντίκτυπο στη ζωή των πολιτών μας. Οπότε, η Υπηρεσία Επικοινωνίας του Κοινοβουλίου έχει αναπτύξει διαφορούς πόρους για να σας βοηθήσει. Παραδείγματο χάρη, το σεμινάριο μεταδίδεται στο διαδίκτυο, οπότε μπορεί να παρακολουθεί κανείς οπουδήποτε υπάρχει ένα Twitter wall και το hashtag είναι EP on migration. Μπορείτε να γράψετε τις απόψεις, να κάνετε ερωτήσεις. Έχουμε ετοιμάσει και ένα βιντεάκι για τις απόψεις των Ευρωπαίων πολιτών, παραγωγή του EPTV, της διαδικτυακής τηλεόρασης του Κοινοβουλίου. Μπορείτε να δείτε αργότερα και μπορείτε ελεύθερα να δημοσιεύσετε στις σελίδες σας μετά από το σεμινάριο. Θα φτιάξουμε και ένα βίντεο για το σεμινάριο αυτό μαζί με κάποιο υλικό στην οπτικοακουστική σελίδα μας το οποίο επίσης θα σας ε, στείλουμε. Θα ήθελα επίσης να τονίσω πως έχουμε διερμηνία σε 8 γλώσσες μεταξύ των οποίων και τα ελληνικά. Η γλώσσα είναι αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ισπανικά, ιταλικά, πορτογαλικά, σουηδικά και ελληνικά. Πολλά τηλεοπτικά και τηλεοπτική και ραδιοφωνική σταθμή εκμεταλλεύτηκαν ευκαιρία για να κάνουν διάφορες συνεντεύξεις για το θέμα. Ελπίζουμε λοιπόν να βρείτε ενδιαφέρον το σεμινάριο. Και τέλος να θυμάστε πως ε, το προσωπικό της μονάδας μας είναι στην διάθεσή σας για να σας βοηθήσει με οτιδήποτε χρειαστείτε. Οπότε, αυτή την ε, στιγμή, ο αρμόδιος ε, συνάδελφος ή αρμόδια συνάδελφος, η Ιζαμπέλ, θα σας εξηγήσει την δουλειά που κάνει το Κοινοβούλιο στους τομείς αυτούς. Ιζαμπέλ, έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ. Καλημέρα σε όλους. Καλώς ορίσατε στο Κοινοβούλιο. Όπως ο Γιάννης σας ανέφερε, εργάζομαι στο υπηρεσία τύπου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και έχω αναλάβει την παρακολούθηση της Επιτροπής των Κοινωνικών Πολιτικών Ελευθεριών και Δικαιοσύνης. Θα σας δώσω μια σύντομη εικόνα για τα βασικά ζητήματα με τα οποία ασχολήθηκε η Επιτροπή αυτή στο παρελθόν και με ποια ακριβώς ασχολείται αυτή τη στιγμή. Οι περισσότεροι ευρωβουλευτές που θα συναντήσετε σήμερα στις 10 και 4 είναι μέλη αυτής της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών και Δικαιοσύνης και είναι οι κύριοι για, τα τρέχοντα ε, θέματα στην διαδικασία συνομοθέτησης με το, με το Συμβούλιο. Δηλαδή το Ευρωκοινοβούλιο νομοθετεί επίσης όρις με τις εθνικές κυβερνήσεις όσον αφορά τις πολιτικές μετανάστευση και ασύλου. Καταρχήν να σας αναφέρω τι έχει κάνει το Κοινοβούλιο σε αυτά τους τομείς. Ήδη έχουμε συντάξει νομοθεσίες περί ασύλου. Ε, το δέσμη για το άσυλο όπως αποκαλείται το 2013 και οι κύριες ε, νομοθεσίες αρχίζουν να ισχύουν από φέτος. Έχουμε δηλαδή τους όρους υποδοχής, έχουμε τη σχετική οδηγία. Πρόκειται για την οδηγία σε ευρωπαϊκό επίπεδο που ασχολείται με τον τρόπο με τον οποίο τα κράτη-μέλη θα πρέπει να υποδέχονται τους ετούντες άσυλο να αναφέρουν υπό ποιες προϋποθέσεις μπορεί αυτοί να κρατηθούν ή όχι. Θα θυμάστε τις πρόσφατες δηλώσεις διαφόρων πολιτικών. Επίσης πρόκειται για την οδηγία που αναφέρει ότι οι μη, τα, μη συνοδευόμενοι ανήλικοι δεν θα πρέπει να περνάνε από κράτηση παρά μόνο σε εξαιρετικές περιστάσεις. Είναι λοιπόν ε, μία από τις βασικότερες νομοθεσίες σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Έχουμε πει την οδηγία με τις διαδικασίες ασύλου. Ένας από τους εισηγητές που θα συναντήσετε σε λίγο είναι η κυρία Σέλβι Κιγιόν που διατέλεσε συντάκτρια της ε, έκθεσης για την οδηγία αυτή και τώρα ε, ασχολείται με την οδηγία για τις τη θέσπιση ενός καταλόγου ασφαλών χωρών προέλευσης. Η οδηγία αυτή χρησιμοποιείται όταν ζητούν άσυλο στην ίδια τους τη χώρα, τη χρονική περίοδο, τους όρους που πρέπει να τηρούνται κτλ. Ένα άλλο, ένα άλλο θέμα είναι το, ο κανονισμός του Δουβλίνου που ορίζει ποιο κράτος μέλος είναι υπεύθυνο για την ε, διεκπαιρέωση της αίτησης ασύλου. Η Κομισιόν ανακοίνωσε ότι ο κανονισμός του Δουβλίνου θα αναθεωρηθεί του χρόνου. Αναμένουμε λοιπόν παρουσίαση πρότασης για αναθεώρηση τον Μάρτιο του επόμενου έτους λόγω των προβλημάτων στην εφαρμογή αυτών των κανόνων. Έχουμε και την έκθεση, τον κανονισμό Eurodac για τα δακτυλικά αποτυπώματα των των άσυλο. Πρόκειται για τη βάση δεδομένων των ετούντων άσυλο που εισέρχονται στην Ένωση και έχουμε και την οδηγία για ε, την χορήγηση διεθνούς προστασίας για κάποιον ο οποίος ε, φεύγει από τον πόλεμο ή τις διώξεις στη χώρα του. Όλα αυτά ξεκίνησαν στην Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών που την οποία εγώ καλύπτω και εγκρίθηκαν από ολόκληρο το Κοινοβούλιο τον Ιούνιο του 2013. Η Επιτροπή και το Κοινοβούλιο επίσης νομοθετούν για τον κανονισμό Frontex. Ξέρετε πως είναι ο οργανισμός που ασχολείται με τα εξωτερικά σύνορα της Ένωσης. Αυτός ο κανονισμός υιοθετήθηκε το 2011 και επίσης πρόκειται να αναφερθεί μέσα μάλιστα σε αυτό το μήνα όπου η Κομισιόν καταθέτει πρόταση για την αναθεώρηση της εντολής αυτού του οργανισμού μάλιστα την επόμενη εβδομάδα. Και επίσης κάτι που ε, αφορά την ε, ομαδοποίηση της ε, συνοριοφυλακής και της ακτοφυλακής της Ένωσης. Κάτι ακόμα το οποίο ασχολήθηκε η Επιτροπή αυτή ήταν η μεταρρύθμιση του Σέγγεν. Οι κανόνες Σέγγεν άλλαξαν επίση το 2013. Το Κοινοβούλιο συνομοθέτησε εκ νέου με τους υπουργούς για τους όρους υπό τους οποίους η προσωρινή έλεγχοι στα εξωτερικά σύνορα επιτρέπονται για περιορισμένες χρονικές περιόδους, καθώς επίσης και για το πώς θα πρέπει να προστατεύονται τα εξωτερικά σύνορα ε, όταν υπάρχει κατάσταση κρίσης, τι θα πρέπει να κάνουν τα κράτη-μέλη ώστε να εξασφαλίσουν την προστασία των σύνορων. Τώρα, αυτό που απασχολεί την Κομισιόν και αυτό θα είναι και το βασικό θέμα στη συνάντηση με τους, με τους ευρωβουλευτές. Ε, έχουμε δύο μηχανισμούς πήγουσας μετεγκατάστασης για το Σεπτέμβριο. Έχουμε τη μετεγκατάσταση 40.000 ετούντων άσυλο και η δεύτερη για 140 ετούντες άσυλο. Αυτά τώρα είναι στην εφαρμοστική τους φάση όπως γνωρίζετε. Η Επιτροπή των Πολιτικών Ελευθεριών τη Δευτέρα το απόγευμα σε μια συζήτηση με το Frontex και την ΕΑΖΟ για το πώς λειτουργούν τα hot spots στην Ελλάδα και την Ιταλία ε, που μπορείτε να τη δείτε σε βίντεο υπάρχει διαθέσιμο. Μέχρι στιγμής μόνο 140 τούντες άσυλο έχουν μετεγκατασταθεί και γι' αυτό και οι ευρωβουλευτές αμφισβητούν τον τρόπο λειτουργίας των hotspot. Πρέπει να λειτουργήσουν καλύτερα ώστε να ε, ολοκληρωθεί ομαλά η διαδικασία μετεγκατάστασης. Θα συναντήσετε επίσης τον Βρετανό ε, Ευρωβουλευτή Τίμωθη Χίρχοπ για τον, για τον μόνιμο μηχανισμό μετεγκατάστασης που δηλαδή θα θέτει σε εφαρμογή αυτή τη διαδικασία, χωρίς να χρειάζεται να περάσουμε από όλη τη διαδικασία που περάσαμε το Σεπτέμβριο. Κάθε φορά δηλαδή για τον μόνιμο μηχανισμό κατάσταση το Κοινοβούλιο θα έχει την εξουσία, την αρμοδιότητα να συναποφασίζει με το Συμβούλιο των Υπουργών. Για τον κατάλογο ασφαλών χωρών προέλευσης. Αυτό ε, ε, στόχο έχει να επιτρέπει την γρήγορη διεκπαιρέωση των αιτήσεων ασύλου, όταν δηλαδή οι πρόσφυγες οι μετανάστες έρχονται από ασφαλείς χώρες θα πρέπει να διεκπαιρωθούν φυσικά οι αιτήσει τους αλλά θα μπορούσαν να διεκπαιρωθούν πιο γρήγορα Έχουμε και το θέμα της Τουρκίας για το κατά πόσο θα πρέπει ή όχι να θεωρηθεί ασφαλής χώρα. Η Τουρκία την περιέλαβε στον κατάλογο της ως ασφαλή χώρα προέλευσης, αλλά κάποιοι ευρωβουλευτές έχουν αμφιβολίες για το κατά πόσο θα πρέπει να περιληφθεί εκεί ή όχι. Οι συζητήσεις στην Κομισιόν ξεκίνησαν αυτό το μήνα και του χρόνου ένα σχέδιο έκθεσης της Σιλβίκη Γιώμ θα υποβληθεί στην Επιτροπή τον Ιανουάριο ή αρχές Φεβρουαρίου. Αναμένουμε να υποβληθεί μέχρι τα τέλη Ιανουαρίου το σχέδιο έκθεσης. Κάτι που επίσης απασχολεί την Επιτροπή είναι η μη συνοδευόμενοι ανήλικη. Ε, μη συνοδευόμενοι ε, ανήλικοι, συνόδευτοι ανήλικοι. Έχουμε συζήτηση από αυτού και θα είναι ενδιαφέρον να ακούσουμε τη Σιλβίκη Γιώμ τι λέει γι' αυτό, γιατί ήταν η εισηγήτρια για το κανονισμό του Δουβλίνου στο παρελθόν. Ε, άλλα θέματα μπορεί να είναι η νόμιμη μετανάστευση που είναι σημαντικό θέμα για την Επιτροπή. Αυτή τη στιγμή έχουμε όρους για είσοδο για τους ε, φοιτητές και τους ερευνητέ. Ήδη υπάρχει συμφωνία με το Συμβούλιο και η ψηφοφορία θα γίνει του χρόνου εδώ στο Κοινοβούλιο. Αναθεώρηση τους οδηγίας για την μπλε κάρτα προβλέπεται για την επόμενη χρονιά και πάλι αυτή η Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών θα ασχοληθεί με αυτό το θέμα. Η αναθεώρηση των νέων κωδίκων θεωρήσεων οι ανθρωπιστικές θεωρήσεις, δηλαδή σημαίνει ότι οι ετούντες άσυλο μπορούν να έρθουν με ασφαλή τρόπο αν έχουν ανθρωπιστική θεώρηση χωρίς να περνάνε από επικίνδυνα ταξίδια, διαθαλάσσεις ή ξηράς. Ε, άλλη σημαντική έκθεση είναι η έκθεση στρατηγικής πρωτοβουλίας για τη μετανάστευση. Η συγγήτρια είναι η Μπερτα Μετζόλα και η κυρία Κέγκε. Εκεί θα συμπεριληφθούν οι βασικές προτεραιότητες του Ευρωκοινοβουλίου με βράχη και μακροπρόθεσμα στον τομέα της μετανάστευσης και της πολιτικής ασύλου. Αναμένεται ψηφοφορία το Φεβρουάριο και από την Ολομέλεια θα πρέπει να περάσει το Μάρτιο. Αυτά λοιπόν ήθελα να σας δώσω μια γρήγορη εικόνα για τα κύρια θέματα και τώρα ο Γιάννης θα συνεχίσει. Χίλια ευχαριστώ Ισαβέλ για αυτή την εκτενή και εξαντλητική και ενδιαφέρουσα παρουσίαση. Ε, της νομοθεσίας ε, που αυτή τη στιγμή είναι στο προπαρασκευαστικό στάδιο στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Θα παρακαλούσα τώρα την κυρία Μαγκένης από την ύπατη αρμοστία του για τους πρόσφυγες να έρθει εδώ στο Προεδρείο. <clears throat> Καλώς ορίσατε όλοι στις Βρυξέλλες ε, σε αυτό το σεμινάριο τύπου για δημοσιογράφους για τη μετανάστευση και το άσυλο. Ελπίζω να μην σας απογοήτευσε ο καλός καιρός. Εχθές ε, έβρεχε, οπότε είδατε τον καιρό των Βρυξελών. Από κακοκαιρία είστε εντάξει, μπορεί να ξαναφτιάξει ο καιρός. Και μπορούμε και να προχωρήσουμε γιατί έχουμε καθυστερήσει, διότι ήταν πολύ μακρές οι διαδικασίες ελέγχου για την είσοδο στο Κοινοβούλιο. Θα δώσω αμέσω το λόγο στη Σοφή Μαγέννη, που είναι επικεφαλής ε, ε, της ε, αντίστοιχης μονάδας τη ΥΠΑ της Αρμοστία στο ΙΕ για τους πρόσφυγες στις Ε, Ξέρετε ότι η Αρμοστία ασχολείται με τα ανθρώπινα δικαιώματα, τους πρόσφυγες και παρακολουθεί όλα αυτά που συμβαίνουν γύρω μας αυτό τον καιρό. Όπως είπαμε και προηγουμένως, είμαστε αναγκασμένοι να μιλάμε εμεί αγγλικά, αλλά εσεί μπορείτε να μιλάτε σε οκτώ γλώσσε. ευχαριστούμε και του Δερμηνεί για την εξαιρετική δουλειά. Η κυρία Μακένη λοιπόν θα κάνει μια σύντομη παρουσίαση γύρω στο δεκάλεπτο και μετά θα ανοίξει η συζήτηση. Επειδή είστε όλοι δημοσιογράφοι, φαντάζομαι και περιμένω ότι θα έχετε καταπληκτικές ερωτήσεις. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα σε όλους σας. Με πολύ χαρά βρίσκομαι ενώπιό σας και βλέπω και τόσο μεγάλη μαζική προσέλευση που δείχνει και το ενδιαφέρον ε, που δείχνει ο κόσμος στην Ευρώπη και παγκοσμίω για τα θέματα του ασύλου και της μετανάστευσης. Σας ευχαριστώ και για την εισαγωγή. Ε, Εργάζομαι στην ύπατη αρμοστία του ΟΗΕ για τους ε, πρόσφυγες. Υπατός ε, ε, αρμοστής είναι ο Αντώνιο Γκουτέρες, πρώην Πρωθυπουργός της Πορτογαλίας. Εδρεύουμε στη Γενέβη. 9.000 υπαλλήλου έχουμε αυτό τον καιρό. Η συντριπτική τους πλειονότητα εργάζεται ανά τον κόσμο επιτόπου. Η πατερμοστία ε, έχει επιχειρησιακή παρουσία και στην Ευρώπη και στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πολλοί από εσά μπορεί να γνωρίζετε και να έχετε έρθει σε επαφή με τις κατατόπους οργανώσεις και γραφεία μας. Ε, ιδρυθήκαμε το 1951 ε, με την αντίστοιχη σύμβαση και το καθεστώ τους μας δίνει τη δυνατότητα και την εντολή να προστατεύουμε τους πρόσφυγες, τους ετούντες άσυλο. Οι ετούντες άσυλο είναι εκείνοι που ζητούν διεθνή προστασία εσωτερικά εκτοπισμένους. Αυτοί είναι άνθρωποι που έχουν εκτοπιστεί εντός των συνόρων της χώρας τους και ε, τους απάτριδες. Απάτριδες είναι εκείνοι που δεν αναγνωρίζονται ως υπήκοοι πολίτες καμιάς χώρας είναι ε, διάφορες ομάδες που εργάζονται εκεί και στο ευρύτερο ευρωπαϊκό πλαίσιο είπατε η αρμοστία του για τους πρόσφυγες έχει κάνει ανθρωπιστική βοήθεια γενικότερα για να προσπαθήσει να αντιμετωπίσει την επίγουσα κατάσταση που βλέπουμε τώρα. Πριν πούμε στην κατάσταση στην Ευρώπη, γιατί φαντάζομαι ότι σε αυτό θέλουμε να εστιάσουμε, γιατί σας ενδιαφέρει ιδιαίτερα, ε, πολύ γρήγορα να σας πω για το παγκόσμιο πλαίσιο. Φαντάζομαι οι ερωτήσεις και απαντήσεις για εσάς στη συζήτηση θα είναι πιο ενδιαφέρουσα από τις παρουσιάσεις. Πώς έχει γενική εικόνα λοιπόν παγκόσμια. Υπάρχει ακόμα η αντίληψη ότι στην Ευρώπη έρχονται οι περισσότεροι μετανάστες, η συντριπτική τους πλειονότητα. Όμως οι στατιστικές αυτού το διαψεύδουν. 8-9 στους 10 πρόσφυγες στον κόσμο, 86% είναι σαν να ε, ε, βρίσκουν υποδοχή στις ε, αναπτυσσόμενες χώρες, όχι στη βιομηχανοποιημένη Δύση. Όταν ο κόσμος αναγκάζεται να βγει στην προσφυγιά, πάει συνήθως στη διπλανή χώρα και ζητάει προστασία. Και τι είδαμε το τελευταίο διάστημα, την τελευταία πενταετία. Είναι πάρα πολλές οι καταστάσεις στον πόλεμο, κεντροαφρικανική δημοκρατία, Μάλι, Λιβύη, βορειοδυτική, βορειοανατολική συγγνώμη, Νιγηρία κτλ. Ε, και πολλές από τις συγκρούσεις αυτές έρχονται να προσθεθούν σε παλαιότερες σειράξεις που δεν έχουν τελειώσει. Το αποτέλεσμα λοιπόν είναι ότι έχουμε μια τεράστια παγκόσμια σύραξη και είναι 16 εκατομμύρια οι ε, εκτοπισμένοι, οι πρόσφυγες. Είναι πάρα πολύ ψηλή αριθμή και είπατε αρμοστία έχει κρούσει τον κόδωνα του κινδύνου. Πρέπει να βρεθούν παγκόσμιες λύσεις γιατί το πρόβλημα είναι παγκόσμιο βασικές χώρες ασύλου, δηλαδή χώρες που υποδέχονται ε, πρόσφυγες είναι η Τουρκία, το Πακιστάν, ο Λίβανος, το Ιράν, η Αιθιοπία και η Ορδανία. Τώρα βέβαια έρχονται ε, πάρα πολλοί σε ορισμένα κράτη-μέλη της Ένωσης, αλλά στη συντεπτική τους πλειονότητα αυτοί βρίσκονται σε χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ας δούμε λοιπόν τι γίνεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Eurostat, που είναι η στατιστική υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δίνει τα στοιχεία για τους ετούντες άσυλο. Κατά το πρώτο τρίμηνο του 2015 ήταν πάνω από 200.000 εκείνοι που ζήτησαν για πρώτη φορά άσυλο και ήρθαν για πρώτη φορά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Από την αρχή του έτους μέχρι τον Οκτώβριο συνολικά πάνω από 800.000 άνθρωποι ζήτησαν άσυλο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Απαντώντας λοιπόν σε κάποιες από ε, αυτές τις αφήξεις και τις απελπιστικές ε, εικόνες που βλέπουμε στη Μεσόγειο, από την κεντρική Μεσόγειο το καλοκαίρι μέσω Ιταλίας και τώρα συνεχίζεται η άλλη οδός από τη Μεσόγειο, από την Τουρκία προς την Ελλάδα. Τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και τα κράτη-μέλη προσπάθησαν να ανταποκριθούν. Ξέρετε, θα ακούσετε μερικά στοιχεία και από τους ευρωβουλευτές, αφού σας κάνω εγώ μια σύντομη παρουσίαση. Δεν θέλω να επιμείνω πάρα πολύ στα μέτρα που ελήφθησαν. Απαντώντας λοιπόν, για να ανταποκριθούμε στις αφήξεις, υπάρχει διαδικασία επανεγκατάστασης και άλλες ε, διαδικασίες ε, που αρχίζουν. Η αρμοστία του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες φρονεί ότι είναι διαχειρίσιμη αυτή η κρίση αν ισχύσουν τα απαραίτητα μέτρα και απαραίτητη αλληλεγγύη που είναι αναγκαία μεταξύ όλων των κρατών μελών. Υπάρχει δυνατότητα αντιμετώπισης. Τι συμβαίνει όμως. Το Ευρωπαϊκό Θεματολόγιο για τη Μετανάστευση έχει διάφορα μέτρα που έχουν ε, ανακοινωθεί ε, για έρευνα και διάσωση για τα hot spots στην Ελλάδα και στην Ιταλία, τα κέντρα καταγραφής που θα διευκολύνουν την επανεγκατάσταση από την Ελλάδα και την Ιταλία και αλλού και σε άλλα κράτη-μέλη. Όλα αυτά ε, υπάρχουν για 20.000 επανεγκατάσταση στην Ευρωπαϊκή Ένωση από γειτονικέ χώρες και επίσης επιπλέον χρηματοδότηση για ανθρώπους που βρίσκονται στην περιοχή για να μπορέσει να σταθεροποιηθεί η κατάστασή τους. Οι πιο πρόσφατες εξελίξεις που μπορεί να τις έχετε παρακολουθήσει κι εσείς, ποιες είναι. Συνεδρίασαν σε σύνοδο κορυφής ε, στις 25 Οκτωβρίου οι ηγέτες ε, των Δυτικών Βαλκανίων και ε, των χωρών που συνιστούν το διάδρομο αυτό και αποφασίστηκε σειρά μέτρων σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μεταξύ των μέτρων αυτών που συμφωνήθηκαν ήταν ότι όλα τα κράτη-μέλη θα συνεργαστούν στενότατα για τη διαχείριση ε, του περάσματος και τη διάφαση μέσω του Βαλκανικού διαδρόμου, έτσι ώστε όσοι χρειάζονται προστασία να έχουν πρόσβαση σε αυτή. Επίσης συμφωνήθηκε να δημιουργηθούν και νέα κέντρα υποδοχής. 50.000 θέσεις στην Ελλάδα και ε, άλλες τόσες στα Δυτικά Βαλκάνια για να σταθεροποιηθεί η κατάσταση και να βοηθηθούν οι άνθρωποι αυτοί που θέλουν να προχωρήσουν, να περάσουν από την Ελλάδα και να ανέβουν προς την ε, Βόρεια Ευρώπη. Ε, πολλά από τα βήματα αυτά είναι στη σωστή κατεύθυνση, αλλά θα πρέπει να γίνουν ακόμα περισσότερα, γιατί η αναγκαία αλληλεγγύη είναι, όπως είπαμε, εκ των όνων ουκάνευ. Στο Λίβανο, στην Ιορδανία και στην Τουρκία πρέπει να σταθεροποιηθεί η κατάσταση. Υπήρξε και σύνοδο κορυφή στις 29 Νοεμβρίου Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας όπου προέκυψαν και κάποιες άλλε συμφωνίες με υποστήριξη και οικονομική τριών δι προ την Τουρκία ε, που θα βοηθήσει τους πρόσφυγες στους οποίους υποδέχεται και φιλοξενεί αυτή τη στιγμή η Τουρκία, κυρίως Σύρους αλλά και από άλλες χώρες. Θέλουμε να τονίσουμε λοιπόν ότι όσο επικίνδυνες και να είναι οι θαλάσσιες οδοί εάν οι οικογένειες δεν έχουν παιδεία, μόρφωση για τα παιδιά τους, δεν έχουν καμιά προοπτική ε, για τη ζωή τους. Ε, δεν βλέπουν τη χώρα τους να βελτιώνεται. Ας πούμε, η κατάσταση στη Συρία, όσο επικίνδυνη και να είναι η κατάσταση, θα προσπαθήσουν να περάσουν αυτή τη θάλασσα, να πάνε πιο πέρα. Θα πρέπει λοιπόν να εξασφαλίσουμε την πρόσβασή τους σε προστασία. Κοιτώ και το χρόνο περίπου έχω ξεπλήσει τα 10 λεπτά, για να προσπαθήσω να σας δώσω μια γεωγραφική εικόνα για το τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή και πόσο επίγουσα είναι η κατάσταση στην Ευρώπη. Βλέπετε εδώ αυτή τη διαφάνεια που ε, αναφέρει τις καθημερινές ημερήσιες αφήξεις στην οδό της Κεντρικής Μεσογείου, τη θαλάσσια οδό που χρησιμοποιήθηκε το καλοκαίρι από τη Βόρεια Αφρική προς την Ιταλία και τη Λαμεντούζα. Αυτή εδώ στο χειμώνα ε, χρησιμοποιείται λιγότερο γιατί είναι ανοιχτή θάλασσα, πέλαγος και δεν είναι δύσκολο να ε, γίνει διάπλους το χειμώνα. Ενώ από την Τουρκία στην Ελλάδα είναι πιο μικρές οι αποστάσεις, μπορεί να είναι λιγότερες οι αφήξεις όταν έχει κακοκαιρία, αλλά συνεχίζουν οι μερίσεις αφήξεις και υποθέτουμε ότι ε, θα συνεχιστούν με αυτό το ρυθμό 4-5 χιλιάδες αφήξεις την ημέρα. Αυτοί οι άνθρωποι θα πρέπει να τύχουν μια υποδοχής και μιας βοήθειας τόπου και ε, στο δρόμο καθοδόν. Και ως αρμόδιος οργανισμός εμείς για τους πρόσφυγες θα πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να δώσουμε ε, βοήθεια στους πιο ευάλωτους και σε εκείνους που πραγματικά ε, αναζητούν προστασία θα πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι αυτές οι ροές είναι κυρίως προσφυγικές. Τα στοιχεία που έχουμε ε, λέγουν ότι πάνω από 80% των ανθρώπων αυτών προέρχονται από εμπόλεμες περιοχές και πάνω από 50% ε, διασχίζουν την, ε, των όσων διασχίζουν τη Μεσόγειο είναι Σύριοι. Δεν χωρά καμία αφιβολία ότι προσπαθούν να ξεφύγουν από ένα τρομακτικό πόλεμο, διώξεις, βία και ένα σωρό δεινά. Από εκεί και πέρα έχουμε πολλούς από το Ιράκ και από το Αφγανιστάν. Δηλαδή είναι κυρίως προσφυγικές αυτές οι ροές. Όλα τα κράτη-μέλη στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν υπογράψει τη Συμφωνία του 1951, τη Σύμβαση για τους Πρόσφυγες και επίσης έχουν δεσμευτεί και έχουν υπογράψει ε, συμβάσεις, θα ακούσετε και άλλα στη συνέχεια, για την προστασία των προσφύγων αυτών. Λοιπόν, ε, είναι τεράστιες οι που υφίστανται και τα κράτη-μέλη και συνεργαζόμαστε μαζί τους έτσι ώστε να ανταποκρίνονται στις υποχρεώσεις τους. Γιατί οι άνθρωποι αυτοί που ζητούν προστασία έχουν δικαιώματα και ε, πρέπει να ανταποκριθούμε σε αυτά. Σταματώ εδώ και θα ακολουθήσει και η συζήτηση. Ναι, ένα χειροκρότημα το αξίζει νομίζω. For sticking... Ιδιαίτερα ε, για την τήρηση του χρόνου. Και τώρα έχετε το λόγο, δεν ξέρω ποιος θέλει. Ε, να σπάσει τον πάγο. Okay. The gentleman over there, please declare your... Παρακαλώ εσείς συστηθείτε, πείτε μας ποιος είστε, από πού είστε, το σύνταγμα που υπηρετείτε και τα λοιπά. Το βαθμό σας και αριθμό μητρό. Uh, uh, my name is Andrea Matisek, I'm from Slovakia. Από τη Σλοβακία Μάτσισεκ λέγομαι, από την Daily Pravda. Είπατε μόλις ότι η πλειονότητα άνω των 80% αν κατάλαβα καλά των ε, αφήξεων είναι άνθρωποι που έρχονται από επόλεμες περιοχές, άρα πρόσφυγες. Είχαμε αυτή τη συζήτηση όμως στην Ευρωπαϊκή Ένωση για το πώς θα διαχωρίσουμε τους οικονομικούς μετανάστες από τους πρόσφυγες. Και δικός μου πρωθυπουργό λέει ότι 80% είπε και 90 μάλιστα ο Πρωθυπουργό μα είναι οικονομικοί μετανάστες. Θα μπορούσατε να μα δώσετε και μια συμβουλή νομική προ μια ευρωπαϊκή κυβέρνηση, προ όλε τι κυβερνήσεις για το πώ θα γίνει ο διαχωρισμός ε, προσφύγων από μετανάστες, γιατί εκεί εστιάζει η συζήτηση σήμερα. Ευχαριστώ. Thank Σας ευχαριστώ πολύ για την ερώτηση. Τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν ήδη καταστήσει διαδικασίες ε, ταυτοποίησης, ε, αναγνώριση εκείνων των ανθρώπων που χρειάζονται διεθνή προστασία. Υπάρχει μια σχετική οδηγία για τις διαδικασίες, ε, για τα πιστοποιητικά. Δηλαδή, όταν έρχεται κάποιος στην Ευρωπαϊκή Ένωση διασχίζει τα σύνορα, φτάνει στα σύνορα και θέλει, θέλω να ο άσυλο, α πούμε, δηλώνει, ε, γίνεται μια αξιολόγηση σύμφωνα με κάποιου κανόνε που είναι γνωστοί και ισχύουν και επιτρέπουν στα κράτη-μέλη να ε, ταυτοποιούν εάν χρειάζεται όντω προστασία ή όχι. Εάν χρειάζεται είτε του χορηγείται το καθεστώ του πρόσφυγα είτε το καθεστώς μια επικουρικής ε, προστασία. Αλλιώς υπάρχει αυτό το καθεστώς ε, ανθρωπιστικής ε, διαμονής ή άλλων ειδών όταν υπάρχει κάποια ιδιαίτερη κατάσταση ε, πιο ευάλωτη και δεν μπορεί να επιστρέψει στη χώρα προέλευσής του. Εάν δεν υπάρχουν άλλοι λόγοι ή άλλο δικαίωμα για λόγους ασύλου προσφυγικού υπάρχει και η διαδικασία για την επιστροφή. Για τον πατρισμό ορισμένο. Ορισμένοι μάλιστα επιλέγουν και εθελοντικά να επιστρέψουν ή άλλοι ε, αναγκάζονται να επαναπατριστούν. Άρα, το θέμα ποιο είναι, να διατηρηθεί ο χώρος προστασίας έτσι ώστε εκείνοι που δικαιούνται προστασίας να έχουν αποτελεσματική πρόσβαση σε αυτή. Ενώ εκείνοι που μπορεί να μην έχουν αυτό το δικαίωμα ή που μπορεί να μην έχουν γενικότερο λόγο να παραμένουν στην Ένωση για λόγους νόμιμης μετανάστευσης ή άλλους ανθρωπιστικούς, τότε θα πρέπει να ε, βοηθούνται εθελοντικά να επιστρέφουν. Έχει πολύ μεγάλη σημασία ιδιαίτερα και για εσά που είστε δημοσιογράφοι η επικοινωνία για αυτό το θέμα. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό, ε, ακόμα και αν είναι πολύ μεγάλα τα νούμερα και οι αφήξεις σε πολλές χώρες ε, κατακλείζουν τα πλήθη, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα πρέπει να υπάρχουν σωστέ διαδικασίε για να ταυτοποιούνται εκείνοι που χρειάζονται προστασία, οπότε αντίστοιχα και εκείνοι που δεν χρειάζονται και δεν μπορούν να έχουν τέτοιε αξιώσει. Το πλαίσιο υπάρχει, αλλά είναι πολλά τα προβλήματα στην εφαρμογή του. Εκεί τα κράτη-μέλη θα πρέπει να συνεργαστούν πάρα πολύ στενά και αλληλέγγυα, έτσι ώστε να μπορέσουν να λειτουργήσουν σωστά αυτές οι διαδικασίες που υπάρχουν. Oui, bonjour, Marianne Meunier du quotidien La Croix. Καλημέρα σας, Μαριάν Μενή, από την ε, καθημερινή εφημερίδα Croix. Μα αναφέρατε διάφορες συμφωνίες που έχουν υπογραφεί από τα κράτη-μέλη της Ένωσης με τρίτες χώρες, αλλά οι επιστροφές πολύ σπάνια γίνονται. Για, γιατί και πώς αντιμετωπίζετε. Yes, it is the case that. Ναι. ναι, όντως. Και το δείχνουν τα στατιστικά στοιχεία. Δηλαδή ο αριθμός όσων επιστρέφουν είναι πολύ χαμηλός. Υπάρχουν επαφές μεταξύ κρατών μελών και άλλων υπηρεσιών για να δούμε πώς θα αντιμετωπιστεί αυτό το ζήτημα. Ίσως είδατε την διάσκεψη της Βαλέτας που ήταν σύνοδος κορυφής όπου οι Ευρωπαίοι ηγέτες και άνθρωποι από τον ΟΗΕ μαζί με τα κράτη-μέλη της Αφρικανικής Ένωσης συναντήθηκαν. για αυτό ακριβώς το ζήτημα, γιατί το όλο ζήτημα των επιστροφών είναι και ζήτημα βορρά-νότου αλλά και μεταξύ των χωρών του νότου. Βεβαίω ε, πίσω από όλα αυτά βρίσκεται η ανάγκη να υπάρξει μια συμφωνία για το πώς θα λειτουργήσουν αυτές οι διαδικασίες ε, και συμφωνίες με χώρες στις οποίες ε, θα επιστρέψουν αυτοί οι άνθρωποι. Γίνονται λοιπόν ε, συζητήσεις για συμφωνίες επανεισδοχής μεταξύ μεμονωμένων κρατών μελών και άλλων κρατών μελών του ΟΗΕ και η Ευρωπαϊκή Ένωση βεβαίω προσπαθεί να δει τι θα κάνει για να λειτουργήσουν τα πράγματα καλύτερα. Από την σκοπιά του ασύλου πρέπει να διασφαλίσουμε πως οι διαδικασίε για την απόδοση προστασίας είναι υψηλή ε, ποιότητας έτσι ώστε να είμαστε σίγουροι ότι όταν τεθεί το ερώτημα το ζήτημα της επιστροφής κάποιου στη χώρα προέλευσής του να είναι σαφές ότι δεν χρειάζεται προστασία ή άλλη ανθρωπιστική βοήθεια. Αυτό ε, είναι κάτι νομίζω το οποίο μπορεί να γίνει για να αυξηθούν οι πιθανότητες επιστροφών. Υπάρχουν και άλλα μέτρα που μπορεί να ακούσετε από άλλες ε, υπηρεσίες ε, στη συζητή σας σήμερα, κυρίως οι εθελοντικοί επαναπατρισμοί. Αυτό φροντίζει ο αδελφός οργανισμός, ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης και είναι κάτι το οποίο κάνουν τα κράτη-μέλη σε συνεργασία με άλλα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα. Αλλά από την δικιά μας τη Σκοπιά βλέπουμε πως μια τέτοια διαδικασία επιστροφών η οποία θα λειτουργεί από τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, είναι σημαντική ακριβώς για να διασφαλιστεί η ακαιρεότητα των συστημάτων ασύλου. Και ένας τρόπος για να βοηθηθεί αυτό είναι να φροντίσουμε να υπάρχει σωστή πρόσβαση σε ποιοτικέ διαδικασίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση Ευχαριστώ. Ραφαέλ Γκοζεντίνα, Ιταλέδη δημοσιογράφος από το Ιταλικό Πρακτορείο Ειδήσεων. Εάν κατάλαβα καλά, ε, είπατε ότι τα hotspot είναι κάτι καλό, γιατί θα γίνει με την κατάσταση των ανθρώπων. Εγώ αυτό κατάλαβα. Στην Ιταλία έχουμε ένα hotspot αυτή τη στιγμή, ε, μια κατάσταση ταυτοποίησης και από αυτό το οποίο βλέπω επιτόπου από τη δουλειά μου είναι το ότι αν η Ιταλία δεχτεί διαχωρισμό μεταξύ οικονομικών μεταναστών και προσφύγων. Κοιτάξτε, εμείς δεν έχουμε Σύριους, έχουμε ανθρώπους από την Αφρική και μέχρι στιγμής με την πολιτική αυτή θα έχουμε μόνο χιλιάδες ανθρώπους χωρίς έγγραφα στη χώρα μας, γιατί θα απορρίπτονται και δεν μπορούν να επαναπατριστούν. Θεωρείται ε, δηλαδή, κατάλαβα καλά, θεωρείτε ότι τα hotspot είναι μια καλή λύση. The idea behind the hotspot. Το σκεπτικό πίσω από τα hotspot είναι να υπάρχει πρόσβαση και προστασία για αυτούς που την χρειάζονται και αλληλεγγύη στην Ιταλία και την Ελλάδα. Ξέρετε πως ε, προφανώς μεγαλύτεροι αριθμοί φτάνουν στον νότο από τις χώρες του Βορρά και ακριβώς ο μηχανισμός ε, μεταγκατάστασης είναι να υπάρχει πρόσβαση άσυλο σε αυτούς που το χρειάζονται αλλά και αλληλεγγύη στην Ιταλία και την Ελλάδα που λαμβάνουν ε, τον μεγαλύτερο αριθμό. Όπως το έχουμε σκεφτεί εμείς ε, και ακόμα βεβαίως είναι νωρίς, υπάρχει μεγάλη πίεση για να αρχίσουν να λειτουργούν πιο αποτελεσματικά Λοιπόν, είναι, έτσι θέλουμε, είναι πως οι ετούντες άσυλο οι οποίοι δέχονται το μηχανισμό μετακατάστασης ε, θα περνάνε από εκεί πέρα μία πρώτη ταυτοποίηση, δακτυλοσκόπηση, θα τους παίρνουν δηλαδή τα δακτυλικά αποτυπώματα και θα Λένε μετά οι άλλες χώρες ε, πως εμείς δεχόμαστε αυτούς τους ανθρώπους ε, να τους πάρουμε από την Ελλάδα ή την Ιταλία αναλόγως. Οπότε τι θα συμβαίνει. Έρχονται οι τούντες ε, άσυλο και η δυνατότητα επεξεργασίας των αιτήσεών τους αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει. Οπότε το σκεπτικό είναι να μεταφέρουμε αυτούς τους αιτούντες άσυλο σε άλλο κράτος της Ένωσης που έχει μικρότερο ποσοστό για να κρυθεί εκεί η υπόθεσή τους. Οπότε θα φύγουν από την Ιταλία ως ετούντες άσυλο χωρίς να έχει κρυθεί ακόμη το εάν δικαιούνται διεθνή προστασία. Θα πάνε σε άλλο κράτος μέλος που θα κρίνει την περίπτωση και αν δικαιούνται διεθνή προστασία θα τους αποδοθεί εκεί. Το κόλπο προφανώς είναι ότι θα πρέπει ο μηχανισμός ε, να μετακινεί ανθρώπους οι οποίοι έχουν πιθανότητα να λάβουν ε, διεθνή προστασία. Δηλαδή να υπάρχει ένας αρχικός έλεγχος για να δούμε ένας άνθρωπος ε, είναι από μια χώρα όπου κανονικά έχει ένα ποσοστό αναγνώρισης προσφύγων 75% και πάνω. Το ποσοστό αυτό είναι το ποσοστό των ανθρώπων ε, από μια χώρα που θεωρούνται πρόσφυγες αφού κρυθεί η υπόθεσή τους. Αυτοί οι άνθρωποι δηλαδή θα μετακατασταθούν από την Ιταλία. Έχουν υπάρξει κάποιες ε, μετακαταστάσεις αλλά πραγματικά αριθμοί είναι πάρα πολύ μικροί. Υπάρχει ένας πίνακας ε, στο site της ε, Ευρωπαϊκής Επιτροπής στη Γενική Διεύθυνση Εσωτερικών και δείχνει πώς δουλεύει ο μηχανισμός. Αλλά καθυστερεί γιατί είναι νέος ο μηχανισμός ακόμα και βεβαίως είναι κάτι το οποίο διαχειρίζονται τα κρατημέλη με τη στήριξη της ε, Frontex και του ΕΑΖΟ, του, της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας ε, Ασύλου. Οπότε επειδή είναι ακόμα νέα η υπόθεση οργανώνεται. Λοιπόν, ο χρόνος πιέζει. Α, τώρα σηκώνεται το χέρι. Λοιπόν, θα ακούσουμε τέσσερις ερωτήσεις, δύο και δύο. Ξεκινήστε από εδώ. Πείτε μας ε, ναι, και παρακαλώ να είστε λίγο σύντομο. Ε, hi, my name is I work for... Ε, Από ένα ισπανικό περιοδικό 5W. Τι κάνει η πατιαρμοστία σε αυτή την κρίση, διότι ε, πολλοί επικρίσεις έχει δεχτεί η Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά η πατιαρμοστία όχι. Έχω πάει σε μέρη που φτάνουν πρόσφυγες Στη Λέσβο, ας πούμε, ε, και δεν είδα κανέναν από την υπατή αρμοστία. Τι κάνει λοιπόν, γιατί όλη την κριτική την ακούει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αν μας άκουγε ο 7χρονος γιος μου, θα ρωτούσε γιατί αφήνουμε τον κόσμο να πνίγεται ή να πληρώνει ε, χιλιάδες δολάρια για να φτάνει στα hot spot στην Ιταλία ή στην Ελλάδα. Γιατί τους αφήνουμε να πνίγονται και να έχουν πληρώσει κιόλα ε, μια περιουσία για να φτάσουν στα hot spots. Γιατί δεν ε, δημιουργούνται τέτοιε δομέ στην Τουρκία, την ίδια ή το Λίβανο. Uh, okay. Μάλιστα. Θα προσπαθήσω να απαντήσω σύντομα. Για να απαντήσω πρώτα στην τελευταία ερώτηση. Τα hot είναι ένα μέτρο μέσα σε, σε ένα πλαίσιο γενική πολιτική και έχετε απόλυτο δίκιο ότι πρέπει να προσπαθήσουμε να δώσουμε ε, βοήθεια και προστασία στον κόσμο πριν κινηθεί. Ε, για να μην πω ότι καταρχήν πρέπει να πάψει αυτή η σύγκρουση στη Συρία που προκαλεί τους πρόσφυγες. Πρώτον και κύριο είναι αυτό. Δεύτερον, ε, όντω πρέπει να στηριχθεί ο κόσμο που βρίσκεται στο Λίβανο και στη Συρία. Πάρα πολλοί κόσμοι από τη Συρία εκεί ζει μέσα σε συνθήκε στόχια. Πρέπει λοιπόν όντω να στηρίξουμε τον αριθμό των καταβλισμών αλλά και να μετακινήσουμε τον κόσμο από αυτές τις χώρες σε ασφαλέστερα μέρη. Τα hotspot λοιπόν είναι τμήμα ευρύτερης πολιτικής και από την άποψη του, της ΥΠΑ της Αρμοστίας θεωρούμε πως από τη στιγμή που συνεχίζεται η σύγκρουση η σύραξη θα κινηθούν και εφόσον κινηθούν θα πρέπει τουλάχιστον να υπάρχει ένα μέρος όπου να μπορούμε να εντοπίσουμε τους πιο ευάλωτους και να τους βάλουμε σε ένα σύστημα που τουλάχιστον να μπορούν να βρουν κάποια βοήθεια. Το θέμα για τη Λέσβο τώρα. Υπάρχει παρουσία στα πέντε νησιά. Έχουμε πολύ προσωπικό που εργάζεται για να στηρίξει και τα hot spot. Δίνουμε πρωτογενή ανθρωπιστική βοήθεια εκεί, μπορούμε να σας δώσουμε τις πληροφορίες για τα πράγματα που προσφέρουμε, κουβέρτες, ε, παλτά, ε, βοήθεια στον κόσμο μόλις φτάνει, έχουμε διερμηνείς, έχουμε κόσμο βοηθά και φτάνει στην Ελλάδα για να έχει πρόσβαση στη hotspot, έχουμε συμβούλους, αλλά σίγουρα δεν αρκούν ε, τα όσα κάνουμε. Δεν υπάρχει αρκετή βοήθεια επιτόπου. Κάνουμε ό,τι μπορούμε, αλλά και πάλι δεν αρκεί. Ευχαριστώ, Σόφη. Λοιπόν, δεν, μπορώ να ακούσουμε, δεν μπορούμε να ακούσουμε άλλες ερωτήσεις, αλλά είμαι βέβαιος ότι η Σόφη με ευχαρίστως θα απαντήσει σε ερωτήσεις σας διμερώς, αν θέλετε. Γιατί έχουμε ένα χρονοδιάγραμμα που καθυστέρησε λόγω των ελέγχων ε, για την είσοδο. Σας ευχαριστώ, εσείς είστε εδώ και θα ζητήσω από τους υπόλοιπους ομιλητές του πρώτου πάνελ να έρθουν εδώ στα έδρανα του Προεδρείου.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 έχουμε τώρα άλλη μια ε, βουλευτή μαζί μας. Λοιπόν, είναι ενδιαφέρουσα η συγκυρία να μιλήσουμε για την ε, μετανάστευση. Να σας πενθυμίσω κάποια πράγματα. Έπρεπε να την είχαμε προβλέψει αυτή την κρίση πριν από τρία-τέσσερα χρόνια, αλλά τελικά η Ευρωπαϊκή Ένωση ανακάλυψε ότι είχαμε πρόβλημα τον Οκτώβριο το 2013 με την ε, τραγωδία της ε, Λαμπεντούζας ε, και τότε ο Μπαρόζο και διάφοροι άλλοι Ευρωπαίοι ηγέτες πήγαν στη Λαμπεντούζα και είπαν όχι πια, αλλά παρόλα αυτά ξανασυνέβησαν αυτά τα πράγματα και τους επόμενους μήνες μέχρι και τον Απρίλιο που μας πέρασε όταν είχαμε πάλι μια νέα τραγωδία στη Λαμπεντούζα η Ιταλία ζήτησε μια Ευρωπαϊκή Σύνοδο κορυφής η οποία τελικά ξύπνησε την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μιλάω για τους ηγέτες ε, περισσότερο παρά για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που το είχε επισημάνει το ζήτημα. Τον Μάιο λοιπόν μετά τη Σύνοδο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε την ε, μεταναστευτική της ατζέντα η οποία πήγαινε πολύ πιο μπροστά από την βούληση των κρατών μελών. Τώρα Βλέπουμε ότι συζητούνται πολλοί νόμοι, γίνονται σύνοδοι κορυφής, ε, ξενυχτάμε στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, αλλά τα αποτελέσματα είναι πενιχρά, γιατί δεν υπάρχει άλλη αλληλεγγύη, δεν υπάρχει επαρκής ε, προστασία στα σύνορα, τα κράτη-μέλη τσακώνονται μεταξύ τους, δεν υπάρχει ενότητα και τελικά ο κόσμος, αν δεν υπάρχουν λύσεις και τελικά ο κόσμος ψηφίζει τη Λεπέν. Οπότε η έλλειψη απαντήσεων από τις ε, κυβερνήσεις είναι το βασικό πρόβλημα που βλέπω εγώ. Ελπίζω λοιπόν να έχουμε την ε, ευκαιρία να ξυπνήσουμε τις ε, κυβερνήσεις και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το ίδιο Λοιπόν, θα αναγνωρίζετε βεβαίως την ε, κυρία εδώ πέρα στα αριστερά μου, την κυρία Σκακέλερ από τους Πράσινους, ήταν υποψήφια για πρόεδρο της Επιτροπής, ε, δεν κέρδισε, αλλά το ξέραμε. Αλλά... Τέλος πάντων ήταν καλή προσπάθεια και πρέπει να ξαναπροσπαθήσετε. Λοιπόν, είναι η συγγήτρια για τον μηχανισμό επανεγκατάστασης. Ε, μετά εδώ πέρα έχουμε την κυρία Σιλβί Γκυγιόμ, σοσιαλίστρια, εισηγήτρια για την, τον κοινό κατάλογο για τις ασφαλείς χώρες προέλευσης όπου δηλαδή αναφέρονται οι χώρες οι οποίες μπορούμε να επαναπατρίσουμε ανθρώπους καθώς θεωρούνται ασφαλείς και βεβαίως έχουμε και τον ε, τον κύριο Χωσέ Μανουέλ Φερνάντες ε, Προσπάθησα να το πω στα πορτοκαλικά. Λοιπόν, έχετε μεταξύ 5 και 10 λεπτών. Ε, ελπίζω να μείνετε στα 5 γιατί ε, οι άνθρωποι αυτοί θα σας, θα γράφουν και εσάς μετά και θα λένε στις ειδήσει, οπότε άμα βαρεθούν θα είναι ανάλογη και η εικόνα σας. Λοιπόν, ξεκινάμε από τις κυρίες. Κυρία Γκυγιόμ. Je vais Ευχαριστώ. Oui, donc... Να βγάλω τα ακουστικά μου. Θα ήθελα να σας πω δύο λόγια για την οδηγία ε, στην οποία θα εργαστώ από τώρα. Στο εξή είναι μια οδηγία Τη οποία η πρόταση κατατέθηκε ε, το Σεπτέμβριο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και είναι μια λογική συνέχεια της δουλειά που είχε ήδη γίνει στην προηγούμενη θητεία για την οδηγία για τις απαιτήσει και τις διαδικασίες του ασύλου. Ήμουν και τότε εισηγήτρια, υπάρχει λοιπόν κάποια συνέχεια στα πράγματα. Άρα λοιπόν ε, γίνεται λόγος για την ασφαλή χώρα καταγωγής, η προέλευση. Θα σας πω τι είναι αυτό για να εννοούμε τα ίδια πράγματα όταν συζητάμε και χρειάζεται αυτό να το διευκρινίσουμε γιατί γίνεται λόγος για ασφαλή χώρα ε, καταγωγής και σε πολλές ε, ε, καταστάσεις και σε πολλά έγγραφα βλέπω να γίνεται λόγος για ασφαλείς τρίτες χώρες. Δεν είναι το ίδιο πράγμα, να το ξεκαθαρίσουμε. Τι είναι λοιπόν η ασφαλής χώρα καταγωγής. Το έχει κωδικοποιήσει η οδηγία για τις διαδικασίες και σύμφωνα με το κείμενο αυτό, μία χώρα θεωρείται ασφαλής όταν έχει δημοκρατικό σύστημα που λειτουργεί με τρόπο βιώσιμο και διαρκή δεν υπάρχουν ε, διώξεις, δεν υπάρχουν απειλές βίας, δεν υπάρχουν εμπόλεμες σειράξεις, ούτε βασανιστήρια, ε, ούτε απάνθρωπες ή εξευτελιστικές ε, τιμωρίες που να επιβάλλονται στον κόσμο. Άρα, όταν κάποιο κατάγεται από αυτή τη χώρα θεωρείται ότι είναι σε ασφάλεια στη χώρα του, οπότε δεν έχει ανάγκη διεθνού προστασία, την οποία ζητεί. Θα καταλαβαίνετε τώρα ότι κατά κάποιο τρόπο ο στόχος είναι να καταπολεμήσουμε τις καταχρήσει ή να ανάρμωστε ή την ανάρμοστη ε, χειραγώγηση ε, της διαδικασίας ασύλου. Πώς ορίζεται μια χώρα ή περισσότερες ως ασφαλείς χώρες καταγωγής. Είναι πολύ σημαντικό αυτό γιατί έχει ε, αυτό συνέπειες και για τις χώρες από τις οποίες ζητείται διεθνής προστασία αλλά και για τους ίδιους τους ετούντες άσυλο. Και να διευκρινίσω κάτι δεν είναι αυτόματο. Όταν κατάγεσαι από μια ασφαλή χώρα δεν σημαίνει ότι δεν έχεις δικαίωμα να ζητήσεις άσυλο, ούτε ότι δεν θα εξεταστεί το έτοιμά σου. Θα τα λέει αυτά και η οδηγία. Και κάθε φορά δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί αυτό ως πρόσφατη ή ως εμπόδιο επειδή κάποιος κατάγεται από μια ασφαλή χώρα. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό να το διευκρινίσουμε. Δεύτερο, που θέλω να ξεκαθαρίσω. Έγιναν επανειλημμένα απόπειρε να ε, γίνει ένας ευρωπαϊκός κατάλογος ε, ασφαλών χωρών. Το είχαμε κάνει και στην οδηγία για τις διαδικασίες για να εναρμονιστεί κάπως η οδηγία αυτή. Να μην υπάρχουν εθνικές λίστες οι οποίες υφίστανται αυτή τη στιγμή στα διάφορα κράτη-μέλη για τις ασφαλείς χώρες. Αυτό δεν κατέστη δυνατό και μετά τις διαπραγματεύσεις εγκαταλείφθηκε. Προς το παρόν λοιπόν συνεπάρχουν διάφοροι εθνικοί κατάλογοι για τις ασφαλείς χώρες ε, καταγωγής και θέλουμε κάπως αυτό να το συντονίσουμε. Επίσης θα πρέπει να κατανοήσουμε σε σχέση με το κείμενο της οδηγίας αυτής ότι οι ροές ε, οι προσεγγίσεις και η διπλωματική στάση κάθε χώρας δεν είναι εναρμονισμένες. Γι' αυτό δεν καταφέραμε να έχουμε μια κοινή ευρωπαϊκή λίστα. Για να σας δώσω κάποια αριθμητικά στοιχεία και να μην μακρηγορώ. 12 είναι οι χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχουν εθνικές λίστες με διαφορετικό ε, τρόπο που έχουν συνταχθεί και διαφορετικό μήκος ε, και διαφορετικό αριθμό χωρών και διαφορετική ακόμα και αντίληψη για την κατάσταση, για το κατά πόσο είναι μια χώρα ασφαλής ή όχι. Παράδειγμα, για κάποιες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Γκάνα θεωρείται, ας πούμε παίρνω μια άλλη χώρα, θεωρείται ασφαλής. Ενώ κάποιες άλλες χώρες της ευρωπαικης ενωσης η γκανα θεωρειται α πουμε παιρνω μια αλλη θεωρούν την Γκάνα ασφαλή χώρα, αλλά μόνο για τους άνδρες. Καταλαβαίνετε πόσες διαφορές υπάρχουν και πόσο δίστανται οι σε αυτό το νομοθετικό λοιπόν κείμενο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι πάρα πολύ ευσύνοπτη πρόταση και ένα παράρτημα με ένα κοινό κατάλογο ασφαλών χωρών καταγωγής Αλβανία, Βοσνία, Ερζεγοβίνη, ε, ε Κόσοβο, Μαυροβούνιο, Σερβία και Τουρκία θεωρούνται ασφαλείς χώρες. Και για να επανέλθω σε αυτό που είχα πει στην αρχή. Τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να ε, διεκπεραιώνουν πιο γρήγορα τις διαδικασίες χορήγησης ασύλου και να υπάρχει και πιο ε, γρήγορη διαδικασία προσφυγής, αν καταλήγουν οι χώρες ότι δεν υπάρχει λόγος διεθνούς προστασίας. Αυτά για να ξεκαθαρίσουμε τις έννοιες και τις πρακτικές προς το παρόν για το συγκεκριμένο κείμενο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Γκυγιόμ. Θα δώσω τώρα το λόγο στην κυρία Σεσίλια ε, Βίξτρομ από τη Σουηδία, φιλελεύθερη ε, και εισηγήτρια για τις αλλαγές στον κανονισμό του Δουβλίνου. Αυτό και αν είναι καυτό θέμα αυτή τη στιγμή. Διότι όπως γνωρίζετε ο κανονισμός του Δουβλίνου ε, προβλέπει ότι η διαδικασία διεκπαιρέωσης τέτοις ενός μετανάστη είναι θέμα τη χώρα στην οποία φτάνει, στην οποία εισέρχεται για πρώτη φορά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αν κάποιο φτάνει από την Τουρκία, αυτή την ευθύνη την έχει η Ελλάδα. Αν φτάνει από τη Λιβύη, την έχει η Ιταλία. Αλλά όταν τόσο μεγάλη αριθμή δεν γίνεται αυτό. Και η Ευρωπαϊκή Ένωση αυτή τη στιγμή με κάποια ε, νοχελικότητα έτσι, συζητάει πώ θα αλλάξει ο κανονισμό του Δουβλίνου, να τροποποιηθεί, ενώ ταυτόχρονα αύριο θα τιμωρήσει κάποια κράτη-μέλη, Κροατία, Μάλτα, Ιταλία και Ελλάδα για ε, ολιγορίες και για παραβίαση του κανόνα για τη δακτυλοσκόπηση. Θα δώσω το λόγο στην κυρία Γουίξτρομ που δυστυχώς θα πρέπει να φύγει γιατί έχει άλλη ενημένη υποχρέωση. Πέντε λεπτά παρακαλώ Σεσίλια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Χαίρομαι που σας συναντώ τέτοια ηλιόλου στη μέρα στις Βρυξέλλες, κάτι το οποίο δεν συμβαίνει συχνά. Έχουμε έρθει να συζητήσουμε εδώ πέρα το κοινό ευρωπαϊκό σύστημα σύλλου. Ήμουν εισηγήτρια, εξακολουθώ να είμαι εισηγήτρια για το Δουβλίνο, καθώς τώρα ασχολούμαστε με τις εξαιρέσεις ε, του κανονισμού του Δουβλίνου, δηλαδή ασυνόδευτους ανηλίκους και την απόφαση του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων που πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη την αναθεώρηση του Δουβλίνου που θα έρθει με μια πρόταση της ε, Κομισιόν τον Μάρτιο όπως ξέρουμε αλλά ήδη από τώρα προσπαθούμε να ευθυγραμμίσουμε τον κανονισμό του Δουβλίνου 3 με την απόφαση του ΔΕΚ. Αν ε, θέλετε διευκρινήσεις ε, να επανέλθω σε αυτό. Λοιπόν, όπως ξέρετε Το κοινό Ευρωπαϊκό Σύστημα Ασύλου αποτελείται από πέντε νομοθετήματα. Η ραχοκοκαλιά είναι το Δουβλίνο, καθώς αποφασίζει ποια χώρα είναι υπεύθυνη για την αξιολόγηση των αιτήσεων ασύλου. Και κατά τη διάρκεια της προηγούμενης θητείας εγκρίναμε έναν αναθεωρημένο κανονισμό του Δουβλίνου. Δυστυχώς πρέπει να πω το Συμβούλιο δεν επέτρεψε κάποια ουσιαστική μεταρρύθμιση του συστήματος, αλλά καταφέραμε να, κάνουμε κάποιες, να επιφέρουμε κάποιες θετικέ αλλαγές όσον αφορά την νομική βεβαιότητα, την εναρμόνιση και την αλληλεγγύη. Ε, κυρίως αλληλεγγύη με τους ε, ανθρώπους, ε, τους ετούντες άσυλο και δεύτερον αλληλεγγύη και μεταξύ των κρατών μελών. Για να ξεκαθαρίσουμε δηλαδή ποιο κράτος μέλος είναι υπεύθυνο και υπό ποιες ε, συνθήκες. Ποια πρέπει να είναι η διαδικασία όταν κάποιος επιστρέφεται στην ε, πρώτη χώρα εισόδου στην Ένωση και έχει πάει σε δεύτερη, τρίτη ή τέταρτη χώρα. Λοιπόν, είναι σαφές σε όλους μας πως το βασικό σύστημα που είχαμε σκεφτεί στο Δουβλίνο δεν λειτουργεί πια. Δηλαδή αν εφαρμοστεί αυστηρά ο κανονισμός ε, του Δουβλίνου υπονοεί πως, ε, και θα σήμαινε πως ο κάθε ένας που μπαίνει στην Ευρώπη θα πρέπει να αξιολογεί από την Ελλάδα ή την Ιταλία. Βεβαίως, αυτό είναι τελείως ανεδαφικό και μη ρεαλιστικό όταν είμαστε 28 χώρες. Επίσης, παράλογο είναι να διακινούνται ελεύθερα τώρα, να ταξιδεύουν ελεύθερα μεταξύ των ε, ευρωπαϊκών ε, χωρών και οι περισσότεροι από αυτούς καταλήγουν σε λίγα κυρίως τη Γερμανία, την Αυστρία και τη Σουηδία όπου καταλήγουν σήμερα το 90% των ετούν τον άσυλο. Και τα δύο αυτά συστήματα είναι εξίσου άδικα. Οπότε η Ευρώπη αυτή τη στιγμή χρειάζεται να μοιραστεί κάπως λογικά τις ευθύνες. Ευθύνες, εμένα δεν μου αρέσει η λέξη βάρος που συχνά γράφουν, γράφεται στα άρθρα σας. Λοιπόν, τις ευθύνες όσον αφορά τους ετούντες άσυλο. Και μάλιστα η Ευρωπαϊκή Ένωση με 500 εκατομμύρια πολίτες και 28 κράτη-μέλη είναι μια πλούσια Ήπειρος, θα μπορούσε, χωρίς ε, σοβαρά προβλήματα, να διαχειριστεί ακόμα και μεγαλύτερες ε, μεταναστευτικές ροές, εάν συντονιστούμε. Δεν μπορούμε να διαχειριστούμε την κατάσταση στα κράτη-μέλη που ανέφερε Γερμανία, Αυστρία και Σουηδία. Έχει ξεφύγει από κάθε έλεγχο η κατάσταση. Το υπογραμμίζω. Γι' αυτό πρέπει να υπάρξει ευρωπαϊκή αλληλεγγύη και να μοιραστούμε τις ευθύνες αυτή τη στιγμή. Και ε, βρισκόμαστε σε μια στιγμή κρίσεως, όχι λόγω της εισρωής. Είναι κρίση ευρωπαϊκής αλληλεγγύης, έλλειψη ευρωπαϊκής αλληλεγγύης. Και βεβαίως τα κράτη-μέλη παίζουν βρώμικα. Λένε ναι θα δε τους δεχτούμε, αλλά όχι στη δικιά μου τη χώρα κάπου αλλού. Και ούτε και σε γειτονική μου χώρα. Οπότε ο κανονισμός ε, Δουβλίνο 3 είναι ένα μέσο του 20ου αιώνα. Είχαμε ξεκινήσει να το συντάσσουμε το 1999. Έχει πλέον ξεπεραστεί. και άρα θα πρέπει να αντικατασταθεί από ένα νέο σύστημα έτσι ώστε να κατανέμονται δικαίως και ισότιμα αιτούντε άσυλο και τα κριτήρια κατανομής πρέπει να είναι αντικειμενικά όπως ο πληθυσμός της κάθε χώρας, το ΑΕΠ της χώρας, το ποσοστό ανεργίας και βεβαίω λαμβάνοντα υπόψη ε, τον αριθμό των άσυλων που έχει υποδεχτεί αυτή η χώρα τα τελευταία χρόνια. Οπότε, δείτε το, δείτε, φανταστείτε την εξή εικόνα. Αν είχαμε παραδείγματο χάρη ένα κομμάτι κεφαλογραβιέρα γεμάτο τρύπε. Αυτό είναι ο οργανισμό του Δουβλίνου. Έχει πάρα πολλέ τρύπε. Γιατί κάθε κράτο μέλος που έχει αναστείλει το Δουβλίνο και αυτό συνέβη πολύ πριν φτάσουμε σε αυτή την κατάσταση. Ε, ήδη τα κρατη είχαν αναστείλει τις επιστροφές ε, στην Ελλάδα πριν από πολλά χρόνια. Μετά από αυτό ανεστάλλει διαδοχικά στη μία χώρα μετά την άλλη. Οπότε έχει καταρρεύσει ουσιαστικά το Δουβλίνο και πρέπει να αντικατασταθεί από κάτι άλλο. Από ένα νομικό μέσο το οποίο θα έχει σχεδιαστεί για τον 21ο αιώνα. Και πραγματικά εγώ αναμένω την πρόταση της ε, Κομισιόν που αναμένεται τον ε, Μάρτιο. Και βεβαίως εμείς ε, θέλουμε να είναι ένα ευρωπαϊκό μέσο. Ευχαριστώ για την προσοχή σας και ζητώ και συγγνώμη που θα φύγω γιατί έχω συνεδρίαση σε άλλη αθουσά, αλλά θα επιστρέψω αν υπάρχει δυνατότητα αργότερα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Βίξτρομ και κύριος Φερνάντες θα μιλήσει τελευταίος γιατί αυτός έχει το χρήμα, είναι εισηγητής ε, για τον προϋπολογισμό. Λοιπόν, να δώσω τώρα τον λόγο στην κυρία Κέλλερ η οποία είναι εισηγητής ε, για το μηχανισμό επανεγκατάστασης που είναι πρόβλημα γιατί αποφασίστηκε το θέμα αυτό. Υπάρχει ένα σχέδιο μετεγκατάστασης μέχρι και 160.000 ατόμων αλλά μέχρι στιγμής ε, έχουν μετακινηθεί 100 με 200 άτομα. Ο πρόεδρος Γιούνκερ είπε ότι με αυτό το ρυθμό θα φτάσουμε την ποσόστοση το 2101 δεν θα είμαστε πια εμείς εδώ. Κάποιος άλλος θα είναι. Λοιπόν, έχετε τον λόγο κυρία Κέλλερ. Σας ευχαριστώ πολύ και ευχαριστώ για την πρόσκληση. Πριν να περάσω στην, με την κατάσταση να πω ο, το πρόβλημα που έχουμε τώρα στην Ευρώπη δεν είναι οι πρόσφυγες. Καταρχήν γιατί ένας άνθρωπος δεν μπορεί να είναι πρόβλημα, ε, αλλά και επειδή ε, ε, δούμε τους αριθμούς, ναι είναι περισσότεροι από ό,τι παλιότερα, αλλά αυτή τη στιγμή έχουμε ας πούμε ένα εκατομμύριο κόσμο που ήρθε φέτος. Που είναι πολύ, ιδιαίτερα αν πάνε μόνο σε ένα-δύο χώρες. Τρεις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν να αντιμετωπίσουν ένα εκατομμύριο πρόσφυγες. Αυτό είναι πολύ. Αν όμως όλες οι χώρες της Ένωσης, 28 κράτη-μέλη με 500 εκατομμύρια κατοίκους απορροφήσουν ένα εκατομμύριο, δεν φαίνονται και τόσοι πολλοί. Και ας μην ξεχνάμε πως άλλες χώρες έχουν πάρει περισσότερους ε, πρόσφυγες. Στην Τουρκία έχουμε πάνω από 2 εκατομμύρια πρόσφυγες. Στο Λίβανο που μόλις 4 εκατομμύρια είναι οι Λιβανέζοι, 1 εκατομμύριο πρόσφυγες έχουν και έχουν ένα, δύο, τρία προβληματάκια περισσότερα. Από ότι εμείς, αν και εμείς το προσπαθούμε να έχουμε λένε και περισσότερα προβλήματα. Άρα λοιπόν το πρόβλημα είναι το να απαντήσουμε στους πρόσφυγες. Εμείς και εκεί λείπει η αλληλεγγύη, όπως είπε και η κυρία Βίξτρομ. Έχουμε βαθιά κρίση στην ευρωπαϊκή αλληλεγγύη, όπως είπε και η Σεσίλια. Ο καθένας θέλει να παίρνει πρόσφυγες, η Ευρώπη, αλλά όχι η χώρα του. Δεν είναι το κοινοβούλιο λοιπόν η Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί εμεί πάντοτε έχουμε πλειοψηφίε και μεταρρύθμιση του συστήματο του Δουβλίνου εδώ και καιρό. Δεν οφείλεται αυτό τόσο στην Κομισιόν, γιατί έχουν ε, υποβάλει μάλιστα φιλόδοξε προτάσει, όλε παραδόξω. Μπορεί να μην συμφωνώ με όλε τι προτάσει του, αλλά εν πάση περιπτώσει, εφόσον έχουν κάνει προτάσει, έχουν και κάποια πολιτική βούληση να δράσουν. Το πρόβλημα είναι τα κάτι μελη που το ένα τα ρίχνει στο άλλο. Ότι εγώ κάνω τα πολλά, ο γείτονά μου δεν κάνει τίποτα και πάει λέγοντα. Και αυτό σημαίνει στην ουσία ότι δεν συμμορφώνονται με την ευρωπαϊκή νομοθεσία που ισχύει. Έχουμε ευρωπαϊκό σύστημα ασύλου. Τώρα μπορεί να πει κανείς ότι δεν είναι αρκετό, δεν είναι καλό, ότι οι ελάχιστε προδιαγραφέ σύμφωνα με του πράσινου δεν αρκούν. Πάντω υπάρχει ένα σύστημα, υπάρχουν προδιαγραφέ. Τα κάτι μέλη όμως δεν το τηρούν και η Κομισιόν ως θεματοφύλακας των συνθηκών δεν έχει ανταποκριθεί στο ρόλο της γιατί μόλις πρόσφατα ξεκίνησε να... κάποιες διαδικασίες κατά παράβαση που είναι καλό αλλά είναι λίγο αργά γιατί εφόσον ε, αν λειτουργούσαν όλα αυτά καλύτερα θα ήμασταν πολύ πιο καλά προετοιμασμένοι και όντως μπορούσαμε να το έχουμε προβλέψει ότι ειδικά οι Σύριοι θα έρχονταν μαζικά φέτος ή εν πάση περιπτώσει ανα πάσα στιγμή γιατί ο πόλεμος εκεί δεν σταματάει επειδή οι γειτονικέ χώρες βρίσκονται σε αυτή την κατάσταση που βρίσκονται και γιατί οι ευρωπαϊκές χώρες ε, ε, δεν έχουν πάντοτε ανταποκριθεί στις θεσμεύσεις τους για το πιστιστικό πρόγραμμα της UNHCR. Και έπειτα υπάρχει και αυτό το θέμα της συνοριοφυλακής. Πολλοί λένε ότι ναι, πρέπει να φυλάσσονται καλύτερα τα σύνορά μας και έτσι δεν θα μπαίνουν οι πρόσφυγες. Μπορεί αυτό να συμβεί αν δούμε την πρακτική στα ευρωπαϊκά σύνορα όπου αποθούνται όντως οι πρόσφυγες, αλλά αν δούμε τη θεωρία και τους νόμους που ισχύουν, που θα έπρεπε να ακολουθούμε, δεν μπορούμε να διώχνουμε τους πρόσφυγες στα σύνορα. Όταν κανείς ζητά άσυλο στα σύνορα πρέπει να τον αφήσουμε να μπει. Οπότε, η ε, φύλαξη των σύνορων δεν θα σταματήσει την εισρωή προσφύγων κανονικά. Μόνο το κλείσιμο και των συνόρων μπορεί να κάνει κάτι τέτοιο και έχουμε αυτό το τεράστιο πρόβλημα ότι ενώ έχουμε σύστημα ασύλου στην Ευρωπαϊκή Ένωση για το οποίο θεωρητικώς είμαστε περήφανοι δεν υπάρχει νομικά πρόσβαση σε αυτό το σύστημα. Περιμένουμε δηλαδή οι πρόσφυγες που θα βρουν προστασία εδώ να βρουν κάποιο παράνομο τρόπο για να μπουν στην Ένωση πράγμα το οποίο είναι γελίο γιατί ο κόσμος πρέπει να μπει σε εκείνες τις βάρκες που βλέπουμε από την Τουρκία προς την Ελλάδα, από τη Λιβύη προς τη Λαμπεντούζα και μετά στην Ιταλία δηλαδή, και στην Ιταλία δηλαδή και αυτές οι βάρκες διαρκώς βουλιάζουν και καθημερινά έχουμε περισσότερους νεκρούς. Μόλις εχθές ακόμα έξι παιδιά πέθαναν στα νυχτά της Τουρκίας των τουρκικών ακτών και καθημερινά συμβαίνει αυτό. Και ε, Μπορεί να μην πεθαίνουν τόσοι πολύ μαζί όπως στη Λαμπεντούζα, αλλά συνεχίζουν καθημερινά να χάνουν τη ζωή τους πολλοί άνθρωποι. Υπάρχει νομική πρόσβαση λοιπόν, όπως στα σύνορα είπαμε. Και ο κώδικας θεωρήσεων προβλέπει η ανθρωπιστική θεώρηση για τον κόσμο που το χρειάζεται, αλλά δεν χρησιμοποιείται. Επίσης έχουμε πρόγραμμα επανεγκατάσταση. Μετεγκατάστασης. Ναι. Με είναι εθελοντικά αυτά τα προγράμματα στα κρατημέλη και δεν τα χρησιμοποιούν συχνά. Γι' αυτό είναι το πρόβλημα που έρχεται ο κόσμος παράνομα και μετά τους τιμωρούμε και από πάνω που έρχονται έτσι παράνομα. Αλλά βασικά δεν έχουν καμία δυνατότητα να έρθουν εδώ νόμιμα. Έχουμε λοιπόν πρόβλημα αλληλεγγύης και ένα μεγάλο κομμάτι αυτού είναι το ε, θέμα της κατανομής. Και εδώ έρχεται η επανεγκατάσταση, γιατί το σύστημα του Δουβλίνου λέει ότι ετούνται σε άσυλο να, κάνουν, να ζητήσουν άσυλο στην είσοδο ε, στην Ένωση, στη χώρα είσοδο. Δεν είναι και πολύ ευφυές αυτό το σύστημα. Και για να ελαφρυνθεί κάπως η επιβάρυνση προς την ε, στην ε, Ελλάδα και την Ιταλία συμφώνησαν τα κράτη-μέλη περίπου να ε, πανεγκαταστήσουν 140.000 κόσμο από 160.000 κόσμο από την Ελλάδα και την Ιταλία. Τώρα οι αφήξεις έχουν μειωθεί λόγω του καιρού και λόγω της συμφωνίας με την Τουρκία. Πάντως αυτό το νούμερο θα είναι γελίο, αλλά ούτε αυτό δεν λειτουργεί. Γιατί τα κράτη-μέλη δεν ανταποκρίνονται σε αυτά που έλαβαν ω υποσχέσει. Δέκα από τη μια χώρα, 30 από την άλλη. Δηλαδή, και πολύ μικρά νούμερα. Είναι υποτίθεται μικρά τα προβλήματα, αλλά δημιουργούν τεράστια προβλήματα για τους πρόσφυγες. Πρέπει να περιμένουν δύο μήνες, ας πούμε, μέχρι να επαναγκατασταθούν. Πώς περιμένετε έναν πρόσφυγα που ζει με τα τελευταία χρήματα που έχει να περιμένει κάπου για δύο μήνες μέχρι ότου ληφθεί απόφαση επανεγκατάστασης χωρίς να ξέρει σε ποια χώρα θα πάει, ούτε αν θα πάει κάπου αλλού. Μικρά εμπόδια δηλαδή υποτίθεται που πρέπει να λυθούν μέχρι ότου να λειτουργήσουν όλα, αλλά και πάλι πρέπει τα κράτη-μέλη να ανταποκριθούν στις ευθύνες τους ε, σοβαρά. Γιατί αλλιώς δεν θα λύσουμε αυτή την κρίση. Την κρίση που όπως είπα είναι κρίση αλληλεγγύης. και περνά και σε πάρα πολλούς άλλους τομείς και νομίζω αυτή είναι η βασική κρίση που έχουμε. Ευχαριστώ. Μάλιστα, πάμε καλά από χρόνο και έχουμε έναν ακόμα μιλητή που μας λείπει, τον Βρετανό Κίρκοπ. Δεν έχει φτάσει ακόμα, αλλά θα φτάσει, μάλλον. Η Σκάκ Κέλλερ ανέφερε το θέμα των χρημάτων και πώς μπορούμε με αυτό να το αντιμετωπίσουμε. Και ο Ευρωπαϊκός προϋπολογισμός μέχρι στιγμής έχει περικοπεί από τα κράτη-μέλη. Ο τελευταίος ήταν ακόμα πιο μικρός από το προηγούμενο και δεν προβλέπονται πολλά χρήματα για τις ευρωπαϊκές πολιτικές διότι οι κυβερνήσεις θεωρούν ότι με αυτόν τον τρόπο μπορείς να πείσεις τους ευρωσκεπτικιστές ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι κάτι που τη δίνεις μόνο λεφτά για να μην κάνει τίποτα. Για την ώρα λοιπόν τώρα η Ευρωπαϊκή Ένωση που πρέπει να δώσει λεφτά δεν έχει. Ο κ. Φερνάνδε που είναι από την Πορτογαλία και από το ΕΛΚ, όπως είπαμε και πριν, το Λαϊκό Κόμμα είναι εισηγητής για το προπολογισμό. Πώς λοιπόν θα βρούμε χρήματα αφού δεν έχουμε. Ευχαριστώ, θα μιλήσω στα πορτογαλικά. Alguns mitos que nós temos em relação ao orçamento. Έχουμε διάφορους μύθους που ισχύουν σε σχέση με τον προπολογισμό και την οικονομία μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ένα, είναι η μεγαλύτερη οικονομία του πλανήτη. Πού ε, και πού το ξεχνάμε αυτό. Και άλλο σημαντικό και ενδιαφέρον στοιχείο είναι ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι το 7% του παγκόσμιου πληθυσμού και ε, κάνει το 50% των κοινωνικών δαπανών στο πλανήτη. Και αυτό το ξεχνάμε. Και ακόμα κάτι. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ο μεγαλύτερος παγκόσμιος δωρητής μέσα σε αυτό το προπολογισμό του 2016 ενισχύσαμε αυτή μας τη θέση και ε, αλλά είναι αλήθεια και αυτό που είπατε, ότι το δημοσιονομικό πλαίσιο 2014-2020 σε σχέση με τα προηγούμενα μειώθηκε, ακόμα και αν υπάρχουν μηχανισμοί ευελιξίας που επιτρέπουν κάποια αντιστάθμιση. Ο προπολογισμό του, του Ευρωπαϊκού, της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, αν θέλουμε να το συγκρίνουμε με τον ομοσπονδιακό ας πούμε προϋπολογισμό των ΙΠΑ είναι 20% του ΑΕΠ αλλά ο δικός μας είναι 1% του ΑΕΠΑ, αλλά έχει μεγάλη προστιθέμενη εξή γιατί το 94% των επενδύσεων είναι δράσεις εμ, ε, και που χρειάζομαστε και περισσότερη ευελιξία και αποφασίσαμε ε, ότι υπάρχει έλλειψη ενός μοντέλου αλληλεγγύης εδώ. Και αυτό, αυτό τα κρατημέλη μεταξύ τους αναλαμβάνουν δεσμεύσεις, τις αναλαμβάνουν, κάνουν μια χαρά ωραίες δηλώσεις, αλλά μετά δεν ανταποκρίνονται σε αυτές. Ενώ εμείς στον προπολογισμό για το 2016 σε σχέση με αυτό το ζήτημα καταρχήν είπαμε ότι οι έκτακτες καταστάσεις θα πρέπει να καλύπτονται από έκτακτα ποσά και ότι δεν μπορούσαμε να μετατρέψουμε αυτούς που είναι θύματα, τους πρόσφυγες, σε ε, θύτες. Γιατί κάποια στιγμή το Συμβούλιο ήθελε να περικόψει πολιτικές, να περικόψει προγράμματα για να μεταφέρει αυτές τις περικοπές σε άλλα προγράμματα, για να βοηθήσει δηλαδή τους πρόσφυγες και να βοηθήσει στα θέματα μετανάστευσης. Αυτή ήταν μια παράδεκτη πρόταση την οποία ποτέ δεν δεχτήκαμε. Και αν κανείς εξετάσει τον προπολογισμό του 2016, αυτές οι κατηγορίες που αφιερώνονται στην ανάπτυξη, στην συνοχή και στην αλληλεγγύη Ε, αυξήθηκαν και για το θέμα των προσφύγων ε, δεν τους εντάξαμε στις κατηγορίες 3 και 4 και χρησιμοποίησαμε κάθε ευελιξία που είχαμε στη διάθεσή μας για να μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε αυτά τα κονδύλια για ώστε να καταπολεμήσουμε την προσφυγική κρίση. Γι' αυτό και πάμε στα όρια, συζητάμε για τα αποθεματικά της κατηγορίας 3 και της κατηγορίας 4 και προσθέσαμε 1,5 δις ευρώ που ήταν το σύνολο του ποσού που υπήρχε στο μέσο ευελιξίας. Για το θέμα της μετανάστευσης και των προσφύγων. Λέγαμε ανέκαθεν ναι, ότι έπρεπε να φτιαχτεί ένα συγκεκριμένο πακέτο για αυτό το στόχο. Είχαμε την εσωτερική αλληλεγγύη και ε, θα πρέπει να έχουμε υπόψη και την εξωτερική αλληλεγγύη. Ένας από τους οργανισμούς επίσης που ασχολούνται με την εσωτερική μας αλληλεγγύη γιατί οι αξίες μας μας επιχρεώνουν να υποδεχτούμε και να ενσωματώσουμε τους πρόσφυγες αλλά και εξωτερική αλληλεγγύη διότι πρέπει να λύσουμε το πρόβλημα στη ρίζα του. Να χρησιμοποιήσουμε κάθε μέσο που έχουμε στη διάθεσή μας για τη συνεργασία και για την ανάπτυξη, έτσι ώστε στην πηγή, στη ρίζα να καταπολεμήσουμε τα αίτια του προβλήματος και να λύσουμε τα προβλήματα της ε, κάθε περιοχής. Δεν είναι τυχαίο, ας πούμε, που ενισχύσαμε την ανθρωπιστική βοήθεια και τη συνιστόσα που απευθύνεται στην εκπαίδευση και την κατάρτιση. 36 εκατομμύρια ευρώ. Αυτή την ενίσχυση τη δώσαμε ότι αυτοί οι νέοι γιατί πάνω από το 50% είναι ε, νέοι που βρίσκονται στα τόπεδα, στα, στους καταβλισμούς προσφύγων, στο Λίβανο, στην Αίγυπτο, στην Τουρκία, στην Ιορδανία. Είναι νέοι άνθρωποι και χρειάζονται ένα σχέδιο για τη ζωή τους. Χρειάζονται αυτή τη βοήθεια που στέλνουμε ώστε να είναι μια πραγματική βοήθεια ε, για να μπορέσουν ε, να έχουν ένα σχέδιο για τη ζωή τους, ένα πρόγραμμα για τη ζωή τους. Στον προϋπολογισμό του 2016, λοιπόν φτιάξαμε ένα πακέτο και πάνω από 10.000 10 ε, δις τα απευθύναμε στην εσωτερική αλληλεγγύη και στην εξωτερική αλληλεγγύη. Είναι προφανές ότι το Ταμείο για το Άσυλο και για την μετανάστευση είναι αυτό που έχει τα περισσότερα χρήματα με 1 δις 200 ε, εκατομμύρια. Έχει μεγαλύτερο βάρος αυτό το ποσό και βοηθά και την ανθρωπιστική βοήθεια που έχουμε το άλλο μεγάλο κονδύλι με άλλο 1,5 δις που βοηθούν και έχουμε επίσης την αναπτυξιακή βοήθεια και το ευρωπαϊκό ε, μέσο γυθνίασης. Τι έκανε λοιπόν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τι έκανε η Κομισιόν για να επιτύχει περισσότερα ποσά, επιπλέον ποσά προχωρη... Ε, ε, συστήσαμε δύο καταπιστεύματα, Trust Funds, το Ταμείο για τη Συρία και το Ταμείο για την Αφρική. Το, αυτό της ε, Συρίας έχει το όνομα Ματάδ και μέσα σε αυτά δώσαμε 3,5 δις. Το Αναπτυξιακό Ταμείο έλεγε έδινε ένα δις και τα κράτη-μέλη θα έπρεπε να συμβάλλουν, να συμπληρώσουν με τα υπόλοιπα χρήματα. Το άλλο καταπίστευμα είναι το Ταμείο για την Αφρική. Για τη Συρία, λέει ο μιλητής, Και πάλι εδώ είχαμε 1,5 δις από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το υπόλοιπο έπρεπε να το συμπληρώσουν τα κρατημέλη. Αλλά τα κρατημέλη βγάζουν λόγους, δίνουν υποσχέσεις και μετά δεν τηρούν αυτές τις υποσχέσεις. Το ίδιο και για το Ταμείο για την Αφρική. Από, τα, από το 1 δις 800 τα κρατημέλη υποσχέθηκαν και έδωσαν 81 εκατομμυριάκια. Δηλαδή λείπουν μόνο 1718 εκατομμύρια ακόμα. Ε, και εκεί στη Συρία υποσχέθηκαν 500, ε, 500 εκατομμύρια ε, και δώσανε 89. Άρα λοιπόν πρέπει τα κατημέλη να σοβαρέψουν λίγο, να ανταποκριθούν σε αυτές τις υποχρεώσεις που ανέλαβαν. Τώρα, για το άλλο ταμείο που λέγεται διευκόλυνση για την Τουρκία όπου θα έχει 3,5 δις. 500 εκατομμύρια θα βγουν από τον προπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα άλλα 2,5 δις πάλι τα κρατημέλη τα υποσχέθηκαν. Εδώ λοιπόν καινοτόμησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τα χρήματα αυτά θα πρέπει να δοθούν πρώτα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και μετά η Ευρωπαϊκή Ένωση θα τα βάλει στην Τουρκία ε, για να υποχρεώσει κατά κάποιο τρόπο η Κομισιόν τα κρατη να ανταποκριθούν στην υποχρέωση που ανέλαβαν. Υπάρχει λοιπόν πέρα από η κρίση της αλληλεγγύης που μόνο επιλύνεται με περισσότερη Ευρώπη, με περισσότερη ε, μοιρασιά, με περισσότερη ε, ε, καινοτομία, αλλά θα πρέπει εδώ ε, τα κράτη-μέλη να ανταποκριθούν και να είναι αξιόπιστα. Όταν λαμβάνουν υποχρεώσεις και μετά δεν τις τηρούν, αυτή η έλλειψη αξιοπιστίας επηρεάζει όλους μας Πάκτα Σουν Σερβάντα θα έπρεπε λοιπόν μέσα σε αυτό το παγκόσμιο, παγκοσμιοποιημένο κόσμο μέσα σε αυτή την κρίση όπου είδαμε να κλείνουν οι πόρτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το αντίθετο θα έπρεπε να συμβαίνει περισσότερη Ευρώπη, περισσότερη ολοκλήρωση με έναν προπολογισμό πιο αλληλέγγυο. Και όχι ο καθένας ε, για τον εαυτό του μόνο και ως όσον εαυτό σωθείτε, γιατί ποτέ δεν πρόκειται να λυθούν τέτοια προβλήματα με αυτόν τον τρόπο. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Φερνάνδες. Ξέρετε, τώρα έχουμε μισή ώρα για ερωτήσεις και απαντήσεις γρήγορες ερωτήσεις. Παρακαλώ να συστήνεστε όνομα, εθνικότητα, ό,τι άλλο έχετε να δηλώσετε. Στο έδρανο 45 παρακαλώ. Και επίσης να μας λέτε και σε ποιον απευθύνετε το ερώτημά σας. Αν αναφέρεστε σε κάποιον συγκεκριμένα. Στο έδρανο υπαριθμό 45, έχετε το λόγο. It's easy. The... The member of the parliament can do it, so you can do it. Μπορούν και οι ευρωβουλευτές να το κάνουν, δεν είναι τόσο δύσκολο, το κάνετε κι εσείς. Πρέπει να είναι εύκολο αφού μέχρι και οι ευρωβουλευτές θα κάνουν. It cannot be difficult. Okay. okay. Ονομάζομαι Γιάννης Ευσταθίου, είμαι Έλληνας δημοσιογράφος από το κανάλι Star. Θα ήθελα να σας ε, επισημάνω το εξής. Ο Βαλκανικός διάβρομος εμποδίζεται για τη διέλευση ε, ανθρώπων που ενδεχομένως και να ζητούν άσυλο από χώρες ε, εκτός από τη Συρία, το Ιράκ και το Αφγανιστάν. Γνωρίζετε όμως ότι μπορεί κάποιος από το Ιράν, μια χώρα που παραβιάζονται τα ανθρώπινα δικαιώματα ή ξέρω εγώ από μια εμπόλεμη περιοχή του Πακιστάν που επίσης κινδυνεύει να είναι βάσιμο, η βάσιμη αίτηση ασύλου. Γνωρίζετε, φαντάζομαι επίσης, ότι ε, πριν από λίγες μέρες έγινε ε, προσπάθεια ε, επιστροφής προσφύγων ή μεταναστών από την Ελλάδα προς το Πακιστάν. Η κυβέρνηση του Πακιστάν δεν επέτρεψε να προσγειωθεί το αεροσκάφο, με αποτέλεσμα να επιστρέψουν πίσω. Με βάση όλα αυτά και με βάση το γεγονό ότι συνεχίζονται οι ροέ αλλοπαπών στην Ελλάδα 3.000-4.000 καθημερινά και ότι από την αρχή του χρόνου έχουν φτάσει περίπου 600.000, δεν είναι βάσιμο ο κίνδυνος εγκλωβισμού εκατοντάδων χιλιάδων προσφύγων και μεταναστών στην Ελλάδα και τι θα γίνει σε αυτή την περίπτωση. Ευχαριστώ πολύ. Ωραία. Και άλλη ερώτηση για να τις ομαδοποιούμε. Παρακαλώ, το όνομά σας, εθνικότητά σας και αμέσως την ερώτηση. Στο έδρανο 79. Ευχαριστώ. Φίλε Ρεν, από μια ισπανική καθημερινή εφημερίδα, το Πούμπλικο. Ε, πορτογαλική, συγγνώμη. Ερώτηση για τη Σκά Ε, μιλήσατε για την ε, επανεγκατάσταση Μα όλα πηγαίνουν τόσο αργά τα πράγματα που οι μη κυβερνητικέ οργανώσεις αρχίζουν να δηλώνουν ότι έχει πεθάνει η πανεκατάσταση πριν καν γεννηθεί. Είναι δηλαδή μια από από αυτή. Εσείς πιστεύετε ακόμα ότι κάποια στιγμή θα αρχίσουν οι χώρες να το υλοποιούν. Είναι ένας μηχανισμός που πριν ε, αφήσει τα πόδια του θα πεθάνει. Ευχαριστώ. Ποιος έχει δικαίωμα στο άσυλο, ποιος θέλει να απαντήσει, εσείς ή η κυρία Κέλλερ. Ναι, παρακαλώ. Ωραία, ευχαριστώ. Η πρώτη ερώτηση δεν ήταν ακριβώς ερώτηση, αλλά πραγματικά υπάρχει ε, κόσμος που έχει μπλοκαριστεί στα Βαλκάνια και με βάση τις εθνικότητες ε, που αυτό δεν συνάδει με τη σύμβαση της Γενέβης, είναι ατομικό το δικαίωμα και εξετάζεται ατομικά η κάθε αίτηση. Δεν μπορεί να πει, ωραία, περάστε οι Σύριοι και καθίστε ε, οι Ιρανοί ή από την Ερυθρέα γιατί έχουν λόγο να ζητούν άσυλο. Όπω και όλα τα 28 κράτη-μέλη πρέπει και η Ελλάδα να κάνει τη δική τη δουλειά. Το μερίδιο που τη αναλογεί. Αλλά είπαμε όλοι ότι θα πρέπει να υπάρξει ένα διαφορετικό σύστημα κατανομή. Προφανώ όχι μόνο η επανεγκατάσταση 160.000 που τώρα έχει αρχίσει. Τι βλέπουμε όλε τι δυσκολίε. Υπήρξαν όμω κάποιε επανεγκαταστάσει Νομίζω έχουμε περάσει τους 200 ήδη και ιδιαίτερα εκείνοι που πήγαν από την Ελλάδα στο Λουξεμβούργο λένε ότι ωραίο που είναι το Λουξεμβούργο και κάνουν και διαφήμιση ε, ε, στην Ελλάδα. Είναι πιο εύκολο τώρα ε, και οι υπόλοιποι να ζητούν επανεγκατάσταση χρειάζεται λίγο καιρό για να στηθεί το σύστημα αυτό και να λειτουργήσει και όταν μπει το νερό στα βλάκια θα είναι πιο γρήγορε οι διαδικασίες. Υπάρχουν ε, μάλλον μικρά αλλά σημαντικά γραφειοκρατικά προβλήματα που πρέπει να λυθούν. Το θέμα είναι τα κράτη-μέλη είναι πρόθυμα να δεχθούν το μερίδιο που τους αναλογεί την ποσόστοση. Εγώ δεν θέλω σε καμία περίπτωση να πω ότι έχει πεθάνει η επανεκατάσταση. Τι κάναμε εμεί πρόσφατα για το άσυλο και τη μετανάστευση ένα θετικό βήμα. Όπως το βλέπω εγώ, τα κράτη-μέλη συμφωνούν ότι πρέπει να στέλνουμε περισσότερους πίσω, περισσότερο έλεγχο των συνόρων, Frontex, μπλοκάρισμα, ε, συμφωνίες με την Τουρκία κτλ. Ενώ η αλληλεγγύη, ε, η υποδοχή των προσφύγων, ε, το μόνο θετικό μέτρο για όλα αυτά ήταν η επανεκατάσταση, 160.000 που αποφασίστηκαν. Εγώ σε καμία περίπτωση δεν θέλω να ε, χαρακτηρίσω γνησιγενή αυτή την προσπάθεια. Αλλά η αρχή, κάθε αρχή και δύσκολη, σιγά σιγά θα βελτιωθεί. Ο κύριος Φερνάντες, για να αρχίσουμε να λύνουμε το πρόβλημα θα πρέπει να πούμε ότι δεν είναι ελληνικό το πρόβλημα. Δεν είναι πρόβλημα της Ελλάδος, είναι πρόβλημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η λύση θα πρέπει να έρθει από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αντί να αντιδρούμε γιατί αυτό κάνει πάντα η Ευρωπαϊκή Ένωση σε όλες τις κρίσεις. Θα πρέπει να δρούμε προληπτικά. Ούτε καλά δεν μίλησα για το ερνηστικό σχέδιο που χρειαζόμαστε για την περιοχή έτσι ώστε ε, να αποφευθούν οι πρόσφυγες. Ε, όλοι συμφωνούμε σε αυτό. Αλλά για να λυθεί το πρόβλημα στη ρίζα του θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν τα κονδύλια. Και δεν μίλησα για ένα ταμείο που είναι εκτός του προπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που θα πρέπει να έχει τον ίδιο στόχο όμως της ανάπτυξης και της συνεργασίας. Αυτό ονομάζεται Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης και για την περίοδο 2014-2020 έχει μια πρικοδότηση πάνω από 31 δισεκατομμύρια ευρώ. Λοιπόν, δεν είναι ελληνικό το πρόβλημα. Ε, όλοι ενεχόμαστε, θα πρέπει να βρούμε λύσεις για τους ανθρώπους αυτούς που βρίσκονται ήδη στα σύνορά μας και έχουμε πόρους γι' αυτό. Ε, βέβαια δεν είναι πολλά τα λεφτά. 6.000 ευρώ ανά πρόσφυγα δίνουμε. Αυτό στον κοινοτικό προϋπολογισμό. Στις μεταφορές δίνουμε 500 ευρώ για τους πρόσφυγες. Έχουμε και άλλα ταμεία για την αλληλεγγύη αυτή. Ας μόνο με τα διαρθρωτικά ταμεία. Και καμιά φορά θα πρέπει να λέμε και το εξή. Υπάρχουν κράτη-μέλη που παίρνουν πολλά χρήματα από την Ευρωπαϊκή Ένωση και μετά δεν είναι σε θέση στην επικράτειά τους να ε, επιδείξουν την απαραίτητη διαλεγγύη. Θα πρέπει να μιλήσουμε και για τα διορθωτικά ταμεία, ιδιαίτερα το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο που μπορεί να βοηθήσει για την ένταξη. Αυτός είναι λοιπόν ο στόχος μας και εντός και των συνόρων, αλλά θα πρέπει οπωσδήποτε να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα και να το λύσουμε εκεί που γεννιέται. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Η συνάδελφος εκεί με το λευκό. Κριστίνα Βίμπερκ ονομάζομαι, είμαι από τη Σουηδία, Ευρωβουλευτής. Ακούτε? Α, μου λέτε ότι δεν είστε δημοσιογράφος. Είστε ευρωβουλευτή. Μα είναι για δημοσιογράφου το σεμινάριο. Αργότερα να κάνετε ερωτήσεις. Όχι ευρωβουλευτέ. Ζητώ συγγνώμη. Θα πρέπει να σεβαστούμε τους κανόνες. Είστε δημοσιογράφος. Ορίστε. Μόνο δημοσιογράφο. Οκ. Τίμα Μπέκ από τη Σλοβακία. Ερώτηση για όλους μάλλον. Όταν μιλάτε για αλληλεγγύη και ότι τα κράτη-μέλη δεν επιδεικνύουν αρκετή αλληλεγγύη, να τα κατονομάσουμε τα κράτη αυτά. Μία από τι χώρε αυτές είναι η δικαιοί μου. Και υπάρχουν και άλλες χώρες που βρίσκονται σε μια κατάσταση τώρα που ε, στη δημόσια συζήτηση ε, μπαίνουν, ε, μπαίνει ένας λόγος της άκρας δεξιάς κατά της Ευρώπης και κατά των μεταναστών και κυριαρχούν αυτές οι διατυπώσεις. Εσείς προσβλέπετε ακόμα στην αλληλεγγύη. Γιατί είπατε ότι υπάρχουν χώρες που παίρνουν χρήματα, αλλά δεν θέλουν να ξέρουν τίποτα μετά για την επανεγκατάσταση. Σας ρωτώ συγκεκριμένα, εσείς τι κάνετε. Υπάρχει ελπίδα αλληλεγγύης. Ζητώ συγγνώμη προηγουμένω μα ρωτήσατε αν είμαστε αισιόδοξοι, επαισιόδοξοι, τώρα αισιόδοξοι. Μα δεν τίθεται έτσι το θέμα. Δεν είναι θέμα αισιοδοξία ή απεσιοδοξία. Εμείς είμαστε προβουλευτές και εργαζόμαστε και έχουμε δεσμευτεί να είμαστε το απαραίτητο αντίβαρο ή ισορροπία απέναντι σε άλλα θεσμικά όργανα. Το είπε πολύ ωραία η απεσιοδοξια εμει ειμαστε προβουλευτε και εργαζομαστε Κέλλερ ότι εμείς λέμε κελλερ οτι εμει λεμε οτι τα κράτη-μέλη δεν ανταποκρίνονται στις υποχρεώσεις τους. Έτσι δουλεύουμε εμείς. Έτσι λειτουργεί το σύστημα. Εμείς θα πρέπει να επιμείνουμε στον υποχρεωτικό χαρακτήρα της ε, κατανομής των προσφύγων. Θα συνεχίσουμε να πιέζουμε. Δεν μας ακολούθησαν. Τώρα τι θέμα αισιοδοξία, αφού βλέπουμε ότι είναι ε, από τους 160.000 έχουν ε, επωφεληθεί 160 άνθρωποι. Τι να πούμε γι' αυτό. Εγώ δεν μπορώ να μιλήσω εξ ονόματο των υπολείπων εδώ συναδέλφων. Η δική μου πρόθεση δεν είναι να ξέρω αν είμαι αισιόδοξη ή απεσιόδοξη. Αυτό δεν έχει σημασία. Σημασία έχει να βρίσκουμε λύσει. Τώρα το πώ το βλέπουν τα κράτη-μέλη. Έχετε δίκιο που αναφέρεστε στη Σλοβακία. Τουλάχιστον ο Πρωθυπουργό χρησιμοποίησε έτσι μια γλώσσα ε, καταδικαστέα. Αλλά και από το δικό μου πολιτικό χώρο ακούγονται τέτοια καταδικαστέα σχόλια. Δεν έχει κανένα δικαιολογίε περισσότερε ή λιγότερε σε σχέση με τον Πρωθυπουργό σα. Η κυρία Σκάκελε. Um, Ευχαριστώ. Να πω πως δεν είναι κάποιες μόνο χώρες που έχουν πρόβλημα με την ελληνική, ούτε καν μόνο οι ανατολικές. Μην έχουμε ένα τεχνητό διχασμό. Παντού υπάρχουν χώρες που δεν ανταποκρίνονται στην αλληλεγγύη. Και βέβαια πάντα εξαρτάται και από το ζήτημα για το οποίο μιλάμε. Συμφωνώ με την Σιλβή, το θέμα είναι τι κάνουμε τώρα, αλλά έλεγα πως είμαι πιο αισιόδοξη για τον κόσμο, ειδικά στην Ανατολική Ευρώπη. Εγώ είμαι από την Ανατολική Γερμανία, όπου είχαμε μεγάλη ιστορία επιφυλάξεων ας πούμε απέναντι στους ξένους γενικώ, αλλά αλλάζει αυτό τα τελευταία 10-15 χρόνια ε, λόγω επαφής ε, με ανθρώπους από άλλες χώρες ε, αλλά και γενικά γινόμαστε πιο ανοιχτοί και πιο σταθεροί στην κατάστασή μας και πολλές ανατολικές χώρες είχαν πολλές ανακατατάξεις στην πρόσφατη ιστορία του. Είμαι λοιπόν αισιόδοξη ότι μπορεί να αλλάξουν τα πράγματα, αλλά χρειάζεται και περισσότερη πολιτική ηγεσία. Δηλαδή ο Πρωθυπουργό πρέπει να πει ότι κοιτάξτε δεν θα είναι εύκολα τα πράγματα, να βοηθήσουμε αυτού του ανθρώπου, θα έχουμε προβλήματα, αλλά είναι άνθρωποι σαν και εσά και εμένα και πρέπει για ανθρωπιστικού λόγου να το κάνουμε. Δυστυχώ βλέπουμε το αντίθετο και πρέπει να πω ότι σοκαρίστηκα από αυτά τα οποία είπε ο πρόεδρος Τούσκ, γιατί ο Τούσκ ως πρόεδρος του Συμβουλίου πρέπει να ενώνει την Ευρώπη και να μην λέει ότι ε, ε, εγώ απ' έξω. Πρέπει να τηρεί και την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Δεν μπορεί να λέει ότι όλα αυτά είναι μπουρδες και πρέπει να σταματήσουμε να δίνουμε άσυλο. Ήταν νομίζω πολύ μεγάλο λάθος. Είναι πάρα πολύ σημαντικό στην Ευρωπαϊκή Ένωση να μην υπάρχει ποτέ διάκριση ανάμεσα σε χώρες που συμβάλλουν αυτές που παίρνουν περισσότερα τις βόρειες χώρες, τις νότιες χώρες, αλλά δυστυχώς ε, πολλές φορές υπάρχουν αυτές οι διακρίσεις, η διχόνοια και σε αυτή την περίπτωση δυστυχώς το ίδιο γίνεται. Για την αλήθεια που υπάρχουν χώρες που παίρνουν πολλά χρήματα από τον προπολογισμό και μετά δεν είναι σε θέση, ζητούν διαρκώς την αλληλεγγύη του ευρωπαϊκού προπολογισμού και παίρνουν ένα σωρό χρήματα και μετά δεν είναι σε θέση να δώσουν μια μικρή βοήθεια και το θέμα που, η ερώτηση που θέσατε δείχνει ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση το θέμα δεν είναι δεξιά ή αριστερά. Έχουμε χώρες όπου κυβερνάει δεξιά που υποδέχονται καλά, ενώ χώρες που κυβερνάει αριστερά και που δεν δέχονται καλά τους ε, ε, πρόσφυγες. Είναι θέμα ηγεσία αυτό. Η Ευρωπαϊκή Ένωση <laughs> πάντα έχει ένα πρόβλημα. Οι εθνικοί ηγέτες τα ρίχνουν όλα τα κακά στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ό,τι καλό κάνουν το διεκδικούν για τον εαυτό τους και πάντοτε αυτό που τους ανησυχεί είναι η κοινή γνώμη. Αν δείτε σε πολλές χώρες θα δείτε ότι τα άκρα αρχίζουν να ε, καταλαμβάνουν τα θέματα και τι κάνουν. Το βλέπουμε και εδώ στο Κοινοβούλιο. Τα άκρα, δεξιά και αριστερά, ψηφίζουν πάντα με τον ίδιο τρόπο. για διαφορετικούς λόγους, ε, αλλά ας πούμε αν μιλήσω για τον προπολογισμό. Πάντα ψηφίσουμε με τον ίδιο τρόπο, η άκρα δεξιά με την άκρα αριστερά. Οι πρόσφυγες είναι θύματα, δεν είναι ένοχοι για κάτι, είναι θύματα των τρομοκρατών και δεν έχουν καμία σχέση με τις ε, τρομοκρατικές επιθέσεις που γίνονται και που έγιναν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουμε μια συλλογική ερώτηση εκεί <laughs> πέρα. Γεια σας από το Σλοβενικό Πρακτορείο Τύπου. Ακούσαμε πολλά χτες και σήμερα για το τι πρέπει να γίνει στην Ευρωπαϊκή Ένωση για να απαντήσουμε σε αυτή την πίεση που βλέπουμε με τους πρόσφυγες, αλλά βλέπετε κάποια αλλαγή στην ζώνη Σέγγεν ως ε, ρεαλιστική πιθανότητα αν δεν γίνουν τα πράγματα όπως πρέπει. Δηλαδή να δημιουργηθεί de facto μία μίνι Σέγγεν ή να ανασταλεί συμμετοχή κάποιων κρατών μελών και για τους τρεις είναι η ερώτηση. Εγώ θα έλεγα ότι αν μπορούσαμε καταρχήν να ε, χρησιμοποιήσουμε όλους τους κανόνες που αφορούν το Σέγγεν πριν να θελήσουμε να του δώσουμε άλλο ρόλο, θα είχαμε ήδη ένα κομμάτι της λύσης. Σίγουρα δεν θα ήταν απόλυτα και ακριβώς αυτό που θα ήθελαν τα κρατημέλη, αλλά πιστεύω πως θα μπορούσαμε ήδη να δούμε κάποιες βελτιώσεις ή αλλαγές, εν περιπτώσει, ε, σε λιγότερο από δύο χρόνια. Προσωπικά και πιστεύω ότι το συμφωνούν με αυτό και η ομάδα μου, δεν υπάρχει ανάγκη να ελέγξουμε το Σέγγεν σε διαφορετικές διαστάσεις, μικρό, μεγάλο, μεσαίο, σε σχέση με αυτό που ισχύει. μάλλον αυτό που χρειάζεται είναι να χρησιμοποιήσουμε το Σέγγεν για το, το λόγο για τον οποίο δημιουργήθηκε, δηλαδή να γίνονται έλεγχοι εξωτερικοί στα σύνορα για να επιτρέπεται μια διάκοπτη ροή στο εσωτερικό. Πράγμα που δεν συμβαίνει τώρα με τα εξωτερικά σύνορα και την υποπτήρια αυτό. Αυτό δεν νομίζω ότι είναι τρελό, αλλά μια μεταρρύθμιση εκβάθρων που θα ξεκινούσε από την αρχή ότι πρώτα πρέπει να φτιάξουμε ένα μεταναστευτικό σύστημα κοινό για ολόκληρη την Ένωση, ένα κοινό σύστημα ασύλου για ολόκληρη την Ένωση και μετά να φτιάξουμε ένα Σέγγεν 2, 3, 4, νομίζω πως δεν είναι καλός δρόμος. Ναι, για την Σέγγεν, ειδικά αυτή η πρόταση των Ολλανδών είναι πολύ ενδιαφέρουσα γιατί θέλουν μια μίνι Σέγγεν για να μας προστατεύσει από όλα τα κακά του εξωκόσμου και μετά συμπεριλαμβάνουν και το Βέλγιο που είναι πάρα πολύ ωραία χώρα αλλά έχει κάποια προβλήματα όσον αφορά την ασφάλεια. Αλλά τέλος πάντων, η Σέγγεν είναι για όλους μας και είναι ένα πράγμα το οποίο είναι απτό για τους πολίτες από την πλευρά της Ευρώπης και δεν θα πρέπει να το θίξουμε και τυχαίνουμε γιατί η Ρουμανία και η Βουλγαρία δεν είναι καν αντικείμενο συζήτησης να μπουν στη Σέγγεν και η πλειοψηφία μπλοκάρει και το συζητάνε τώρα έντονα στο Συμβούλιο δεν είναι καν προσυζήτηση να πω πως ε, για την ε, άκρα δεξιά και άκρα αριστερά μην τα βάζετε αυτά όλα μαζί. Ε, πείτε λαϊκισμό και τα λοιπά, αλλά μία πλευρά μόνο αρνείται ανθρώπινα δικαιώματα στους πρόσφυγες και τα λοιπά. Η αριστερά δεν το κάνει αυτό. Μπορεί να μη συμφωνείτε, αλλά μην μας βάζετε όλους μαζί στο ίδιο τσουβάλι. Ευχαριστώ. Συμφωνώ με τις ε, συναδέλφους. Τώρα, ε, η διάλυση της Σέγγεν σημαίνει διάλυση της Ευρώπης. Βελτιώσεις πάντα χωράνε, ιδιαίτερα ε, για τα εξωτερικά σύνορα. Είναι υποχρέωση των κρατών μελών, αλλά και ολόκληρης της Ευρώπης. είναι και θέμα ασφάλειας που πρέπει να εξασφαλίζουμε για την Ευρώπη. Και αυτό δεν γίνεται ε, διαφορετικά παρά μόνο με ενίσχυση των εξωτερικών μας συνόρων. Εδώ κάποιος εκ δεξιών. Όσο γίνεται πιο ευσύνοπτα. Ευχαριστώ. πάρα πολύ. Να σας ευχαριστήσω όλους σας για αυτά τα οποία είπατε. Το ερώτημά μου αφορά τις αλλαγές ε, στο Δουμπλίνο όπως είπατε θα μεταρρυθμιστεί τον Μάρτιο υπάρχει ένα επίμαχο θέμα που αφορά τον κανόνα για την πρώτη χώρα εισόδου η οποία είναι υπεύθυνη όχι μόνο για την διαδικασία ασύλου αλλά αναλαμβάνει και την ευθύνη για το άτομο αυτό για την παραμονή του στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα ήθελα να μάθω λοιπόν εάν ε, θα παραμείνει αυτό το κομμάτι μετά την μεταρρύθμιση, πώς έχει η κατάσταση για το τμήμα αυτό της νομοθεσίας, πώς έχουν τα πράγματα. Ε, Δεν είναι ακριβώς απάντηση, μάλλον προέκταση της ερώτησής σας. Σας είπαμε τους λόγους προηγουμένως. Γιατί έχει έρθει αυτή η πρόταση κατανομής των ε, μετακινουμένων. Κατά κάποιο τρόπο αυτό αντιστοιχεί σε αναστολή ε, του Δουβλίνου. Η διακοπή. Γιατί ακούσαμε προηγουμένως τη μέθοδο ε, κατανομής. Άρα, de facto, είναι σε διακοπή, αναστολή ο κανονισμός του Δουβλίνου. Γιατί θα πάμε τώρα σε ένα Δουβλίνο 4 πιθανότατα αφού δεν καταφέρνουμε με πολύ μεγάλη δυσκολία για να είμαι αισιόδοξη όπως είπατε προηγουμένως δεν καταφέρνουμε να ολοκληρώσουμε το σύστημα ανακατανομής των ανθρώπων αυτών. Εκεί υπάρχει έλλειμμα, υπάρχει πραγματικό ερωτηματικό. Τι το θέλουμε το νέο σύστημα, γιατί νέα τροποποίηση του κανονισμού Δουβλίνου 3 για να γίνει ένα Δουβλίνο 4. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε λύσει ε, το σύστημα ε, με άλλους τρόπους για την αναδιανομή. Ε, η δικιά μου η πρόβλεψη, τόσο δεν ξέρω τι θα προτείνει η Κομισιόν, γιατί πρέπει να κινηθεί μεταξύ δύο πόλων μάλλον το Κοινοβούλιο θα ζητήσει ένα τελείως διαφορετικό σύστημα που θα προβλέπει μια δίκαιη κατανομή των κρατών μελών. Μάλλον το Συμβούλιο θα διαφωνήσει και μετά θα δούμε τι θα βγει. Και δεν πρέπει να ξεχνάμε πώς μιλάμε για ανθρώπους εδώ πέρα, όχι για πακέτα Γι' αυτό πρέπει να συμπεριληφθούν και οι προτεραιότητες ε, των προσφύγων, π.χ. οικογενειακοί δεσμοί ή αν μιλάνε κάποια γλώσσα κτλ. Αυτό είναι μια σημαντική πτυχή που εμείς οι πράσινοι θα προσπαθήσουμε να προωθήσουμε. Μάλιστα, πέντε λεπτά έχουμε ακόμα. Μπορούμε να ακούσουμε κάποιες ερωτήσεις ε, έτσι γρήγορα. Η κυρία εκεί και μετά ο κύριος εκεί πέρα. Και εγώ από τη Σλοβακία Σλοβακική ραδιοτηλεόραση. Ξέρω πως υπάρχει αυτή η αισιοδοξία, απεσιοδοξία, αλλά ας το δούμε ρεαλιστικά. Σλοβακία ξέρετε πως ε, δεν υπάρχει περίπτωση να δεχτεί. Ξέρετε τι έγινε και την προηγούμενη φορά. Δεν θα επαναλάβω τα επιχειρήματα. Ε, του χρόνου λοιπόν ε, φαντάζεστε θα υπάρχουν ακόμα χώρες σαν την Πολωνία, Σλοβακία, Ουγγαρία που δεν θα δεχτούν πρόσφυγες και κάποιος θα πει, ε, δηλαδή πόσους περισσότερους ε, πρόσφυγες ε, θα πάρουμε, ποιο νούμερο βλέπετε εσείς, μάλιστα. Και εδώ πέρα, κύριος εδώ μπροστά. Αρκεί να μην είστε Σλοβάκος, όχι Πορτογάλος είμαι θα ήθελα να πω το εξή. Ακούσαμε πάρα πολλά. Σήμερα η κρίση αλληλεγγύης ε, είναι κάτι που ακούσαμε. Αλλά απλά έτσι δηλαδή η Ευρωπαϊκή Ένωση κρύβει την έλλειψη στρατηγικής για να αντιμετωπίσει το ζήτημα αυτό. Ε, θα ήθελα να μάθω εάν η Ευρωπαϊκή Ένωση κοιτάει πώς θα σταθεροποιήσει μακροπρόθεσμα τις χώρες αυτές στην Αφρική και τη Μέση Ανατολή για να αντιμετωπίσουν την κλιματική αλλαγή. Έχουμε αρκετά λεφτά να αντιμετωπίσουμε αυτό το ζήτημα και για πώς. Θα ήθελα για να σας δώσω μια ιδέα ε, για τους αριθμούς και τα μεγέθη. Είναι σημαντικό. 60 εκατομμύρια κάθε χρόνο η πρόσφυγες, 60, συγγνώμη, έχει 16, 60 εκατομμύρια το χρόνο ε, μετακινούνται. Στην Ευρώπη είναι απειροελάχιστες ε, οι διαστάσεις σε σχέση με το παγκόσμιο φαινόμενο. Θα πρέπει να δούμε και πώς μετακινούνται πάνω από 80% των ανθρώπων αυτών που είναι αναγκασμένοι να φύγουν από την πατρίδα τους για κάποιο χώρο. Ε, είναι σε γειτονικέ χώρες. Δεν έχουμε μεγάλες μετακινήσεις πληθυσμών, μαζικές ε, νότου προς το βορρά, όπως καμιά φορά υπάρχει αντίληψη. Θα πρέπει να ξέρουμε και πόσοι έχουν φτάσει στην Ιορδανία, στο Λίβανο, στην Τουρκία αν κάνουμε κάποιες προβολές, εγώ είμαι Γαλλίδα, δεν είμαι Πορτογαλίδα, αν το αντιστοιχίσουμε στη Γαλλία, αυτό θα σημαίνει 17 εκατομμύρια σε σχέση με τον πληθυσμό της χώρας. Θα πρέπει να καταλάβουμε για ποια τάξη μεγέθους μιλούμε. Στις χώρες της Ένωσης λέμε ότι είναι ε, πολλοί όσοι φτάνουν, αλλά δεν καταλαβαίνουμε τι σημαίνει αυτό ε, για χώρες που συνιστούν το 1 τρίτο ή το 1 τέταρτο του πληθυσμού τους. Καμιά φορά αντιδρούμε με βάση την επικαιρότητα ή την κοινή γνώμη για τον τρόπο με τον οποίο υποδεχόμαστε και πόσους θα πάρουμε κτλ. Αλλά καμιά φορά να έχουμε υπόψη μας και τα μεγέθη. Και για ποια τάξη μεγέθους μιλάμε. Στρατηγική τώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης αν υπάρχει για αυτά τα θέματα. Ε, Προφανώ δεν υπάρχει ευρωπαϊκή στρατηγική γενική και αόριστη και παγκόσμια. Υπάρχει στρατηγική τη Ευρωπαϊκής Επιτροπή και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Και το περιγράψαμε. Και σύμφωνα με μια αντίληψη που είναι πλειοψηφική. Δηλαδή ότι να δούμε και το κακό επί τόπου στη ρίζα του, να δούμε τι γίνεται με την ένταξη και με νόμιμες οδούς μετανάστευσης. Έχουμε ένα συλλογισμό και μια αντίληψη που νομίζω ότι στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κυριαρχεί. Αυτό μεταφράζεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε παραγωγή κειμένων. Μπορεί τώρα να φαίνονται κάποιες κινήσεις σπασμωδικές, αλλά τα κράτη-μέλη είναι το ζήτημα. Είναι σαφέστατο. Τώρα αν είσαι αισιόδοξο, αποσιόδοξο, το θέμα είναι εάν θα προσεγγίσουν οι θέσεις των κρατών μελών. Εγώ δεν είμαι πυθία για να ξέρω τι θα γίνει, ε, αλλά έτσι πρέπει να διαχειριστούμε την κατάσταση. Όσον αφορά την στρατηγική, κοιτάξτε, νομίζω πως ε, οτιδήποτε κάνουμε είναι καλύτερο από οτιδήποτε κάνει ένα κράτος μέλος. Οπωσδήποτε η αναπτυξιακή συνεργασία είναι ένα τέτοιο θέμα. Ξέρετε, κάθε φορά που βυθίζεται μια βάρκα, ακούω του συναδέλφου στην Ολομέλεια πω πρέπει να κάνουμε κάτι με την αναπτυξιακή συνεργασία. Άμα το θυμόμαστε αυτό, δηλαδή μόνο κάθε φορά για να σταματήσουν οι πρόσφυγε ε, δεν αρκεί. Επίση δεν είναι μόνο λεφτά που στέλνουμε αλλού, είναι και οι πολιτικέ που κάνουμε εδώ πέρα, που ασκούμε εδώ πέρα, που είναι καταστατικέ, όπω ε, η γεωργική εμπορική πολιτική που θα μπορούσε να υποστηρίζει την ανάπτυξη. Πρέπει να αλλάξουμε και κάποια πολιτική μας. Αλλά μετά έχουμε ζητήματα όπως τα γεωργικά συμφέροντα, η αλληλεία στην Πορτογαλία κτλ. Και μετά γίνονται δύσκολα τα πράγματα. Και όταν φτάνουμε σε αυτές τις ψήφους μετά πολλοί συνάδελφοι μετά δεν σκέφτονται την ανάπτυξη άλλων χωρών. Σε ένα χρόνο, ναι, Σίγουρα θα έχουμε χώρες οι οποίες δεν θα υποδέχονται τόσο καλά. Αναμένω να δω τι θα κάνει η Σλοβακία με την Προεδρία. Είμαι περίεργη να δω. Τώρα για το νούμερο. Δεν μπορούμε να βάλουμε ανώτατο όριο στο άσυλο. Γιατί ο κόσμος έχει δικαίωμα να ζητάει άσυλο. Θα διώξουμε τον πρώτο Σύριο μετά το εκατομμύριο και θα του πούμε ότι φτάσαμε στο όριο. Όχι, κανείς μας δεν θα το έκανε αυτό. Και πρέπει να αυξήσουμε την ε, ικανότητα απορρόφησης όσο δεν σταματά ο πόλεμος Συρία και μάλλον δεν γίνεται αυτό και γι' αυτό πρέπει τα κράτη-μέλη να επιδείξουν ε, αλληλεγγύη για αυτή την πάρα πολύ βασική ανθρώπινη ανάγκη. Λοιπόν, να σταματήσουμε τώρα. Θέλετε να πείτε κάτι. Αλλά. Μ' αρέσει όμως να παραβιάζω τους κανόνες. Λοιπόν, θα δώσω τον λόγο για μια πάρα πολύ καλή ερώτηση. Ποιος θα κάνει τέτοια ερώτηση. Λοιπόν, εκεί πέρα προσπαθείτε. Πείτε μου όνομα, από που είστε κτλ. Τι είναι, τόσο δύσκολο είναι. Α, ναι, δουλεύει. Ωραία. Μπάλα από την Ουγγαρία. Δεν... Ε, αλλά εργάζομαι για την Interstandard, την αυστριακή εφημερίδα. Ας υποθέσουμε ότι ξεκινήσει αυτό το σύστημα επαναγκατάστασης και το δεχτούν 28 χώρες και τα λοιπά. Πώς μπορείτε να μας εγγυηθείτε ότι οι πρόσφυγες οι οποίοι θα πάνε σε χώρες όπως Ρουμανία, Βουλγαρία, Ουγγαρία θα παραμείνουν σε αυτές τις χώρες και δεν θα φύγουν εντός 24 ωρών για Γερμανία, Αυστρία και Σουηδία. Ναι, πρώτα απ' όλα διασφαλίζοντας ότι η Ουγγαρία και οποιαδήποτε άλλη χώρα του συμπεριφέρεται σωστά αν τους βάζετε στη φυλακή όπως τώρα δεν είναι έκπληξη ότι δεν θέλει να πάει κανείς στην Ουγγαρία. Δεν θέλουν να πάνε οπωσδήποτε στη Γερμανία και τη Σουηδία, αλλά δεν θέλουν να πάνε στην Ουγγαρία. Έχετε ένα πρόβλημα εικόνας ε, που πρέπει να διορθωθεί. Δεύτερον, μέσω τη πρόληψη. Πρέπει να λάβουμε υπόψη τι προτεραιότητε των προσφύγων. Γιατί αν στείλουμε κάποιον σε μια χώρα ε, παρά τη θέλησή του, γιατί η οικογένειά του είναι αλλού, και εμεί τον στέλνουμε σε άλλη χώρα, ναι, θα πάνε στην άλλη χώρα. Αλλά αν πούμε ναι είναι δυνατόν ότι ε, λυπούμαστε. Δεν είναι δυνατόν αλλά και αυτή η άλλη χώρα ωραία είναι γιατί η γλώσσα είναι παρόμοια ή με τα προσόντα σας τα βρείτε δουλειά κτλ. Και όσο διαρκεί η διαδικασία του ασύλου θα σας κρατήσουμε ή άλλο ένα χρόνο αλλά όχι η όλη αυτή η διαδικασία συν πέντε χρόνια γιατί αυτή μπορεί να διαρκέσει ποιος ξέρει πώς μπορεί να πει ότι εντάξει θα μείνω για αυτό το διάστημα εκεί. Αλλά ε, πρέπει να θυμόμαστε ότι μιλάμε για ανθρώπου και όχι για πακέτα και μπορεί να γίνουν τα πράγματα πολύ καλύτερα από όσο έχουν αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, να ευχαριστήσω τώρα τους ομιλητέ μας, ε, τον κύριο Φερνάντε τη Σβίγκη Γιώμου, τον κύριο Κέλλερ. Δεν ευχαριστώ αυτού που δεν ήρθαν. Ε, και τώρα έχουμε Ακόμα μια ώρα για το επόμενο πάνελ και μετά έχουμε διάλειμμα για φαγητό. Υπομονή λοιπόν. Hello. Are you ready? Είστε έτοιμοι. Now, if Λοιπόν, αν νομίζατε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει πρόβλημα φύλου, ισορροπίας, τώρα είστε βέβαιοι. Έχουμε τέσσερις γυναίκες και έναν άντρα. Τα συμπεράσματα δικά σας. Ποιος έχει το πρόβλημα φύλου. Ε, αλλά εγώ με χαρά το υφίσταμαι όλο αυτό. Δύο ανακοινώσεις. Πρώτον, σας θυμίζω ότι πρέπει να υπογράψετε εδώ στον κατάλογο παρουσιών. Δεν ξέρω για ποιο λόγο, έτσι μου είπαν να σας πω ότι πρέπει να υπογράψετε. Δεύτερον, βλέπω διαφόρους να κυκλοφορούν με iPad, θα τους δείτε κι εσείς, αξιολογούν τη συζήτηση, ρωτάνε και να είστε ευγενικοί μαζί τους. Παρακαλώ. Λοιπόν, πριν σας συστήσω το επόμενο πάνελ, Νομίζω έχουμε ένα πάρα πολύ μικρό σύντομο βίντεο που θα προβληθεί τώρα εάν ε, είναι σωστή και υλοποιείται η υπόσχεση. Το έχουμε έτοιμο το βίντεο. Είναι σύντομο. Crisis reached critical intensity. A survey was conducted in 28 member states with 28,150 citizens above the age of 15.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 μας δείχνει το βίντεο γιατί είμαστε εδώ σήμερα. Έγινε μια δημοσκόπηση από το Ευρωβαρόμετρο που ρώτησαν τους Ευρωπαίους πολίτες τι πιστεύουν για τον δρομοκρατία ε, ε, και τη μετανάστευση. Σωστά είπε η κυρία Βόζεμπερκ, αυτό έγινε ένα μήνα πριν τις επιθέσεις στο Παρίσι και πιθανώς αν ξαναγίνει τώρα οι απαντήσεις θα είναι διαφορετικές, όχι τόσο καλές εν πάση περιπτώσει δηλαδή όχι και πολύ άσχημες, γιατί υπάρχει μια κοινωνική συζήτηση μεταξύ, και συνείδηση μεταξύ των πολιτών που είναι υψηλότερη ίσως από των ηγετών καμιά φορά. Είδατε λοιπόν το Ευρώπα-Μέτρο, έχουμε τέσσερις ευρωβουλευτίνες ε, από κέντρο αριστερά και, πέρα, ε, και είχαν προσκληθεί και από την ομάδα της Λεπέν και από τη Λέγκα ε, και αρνήθηκαν την παρουσία τους. Εντάξει, τι να κάνουμε τώρα. Ε, τέσσερις κυρίες λοιπόν, θα σας συστήσω με τη σειρά. Συνήθως δίνω το λόγο πρώτα στις κυρίες, αλλά αφού έχω τέσσερις αλφαβητικά. Λοιπόν, η κυρία Μπιόρκ θα μιλήσει πρώτη, είναι από την Ενωτική Αριστερά, από τη Σουηδία. Πέντε λεπτά παρακαλώ και μετά ερωτήσεις. Ευχαριστώ, θα μιλήσω σου ειδικά, που έχω την ευκαιρία. Λοιπόν, βάλτε τα ακουστικά σας, ε, σας παρακαλώ. Λάβαμε κάποιες ε, ερωτήσεις ε, πριν από την συνάντηση αυτή και δεν μου κάνει εντύπωση βλέποντας τις ερωτήσεις αυτής, ε, αυτές 60 εκατομμύρια άνθρωποι αυτή τη στιγμή είναι πρόσφυγες όπως είπε η Ίσκα Κέλλερ, οπότε προφανώς χρειάζεται κάποια πολιτική ηγεσία, πρέπει να πάρουμε την υπόθεση αυτή στα σοβαρά, υπεύθυνα, ανησυχώ γιατί βλέπουμε πως οι πολιτικοί ηγέτες κάνουν το αντίθετο. Δημιουργούν φόβο, παίζουν με τον εθνικισμό και είναι και ρατσιστές. Για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Και νομίζω πως το ακριβώς αντίθετο χρειαζόμαστε. Χρειάζεται πολιτική ηγεσία, επικοδομητική για το μέλλον της Ευρώπης, να λάβουμε μεγαλύτερη ευθύνη για τους ανθρώπους αυτούς. Όπως είπαν και άλλοι στο πάνελ, στην Ευρώπη δεχόμαστε μικρό ποσοστό των ανθρώπων αυτών και νομίζω πως είναι πάρα πολύ σημαντικό να μην μπερδεύουμε τα διαφορετικά ζητήματα. Είναι παλιά συνήθεια αυτή, μπερδεύουμε τις πρόσφυγες με τα ζητήματα ασφαλείας, μπερδεύουμε την οικονομική κατάσταση με την έλλειψη Κοινωνική ασφάλεια που αισθάνεται τον κόσμο με το θέμα των προσφύγων. Οι πολιτικοί ηγέτε πρέπει να το δουν το ζήτημα συνολικά. Το θετικό στο φιλμάκι αυτό είναι πως ε, ο κόσμος αντιλαμβάνεται πως χρειαζόμαστε μεγαλύτερη ευθύνη στο ευρωπαϊκό επίπεδο και νομίζω πως ε, χρειάζεται περισσότερη στήριξη από αυτή την οποία βλέπουμε στο Συμβούλιο. Ο κόσμος πρέπει να αντιληφθεί πως η Ευρώπη της ιστορίας δεν είναι... Η ιστορία της Ευρώπης, δεν είναι ενός πολιτισμού μόνο. Δεν υπάρχει μέλλον για την ακροδεξιά πολιτική. Πρέπει να δώσουμε λύσεις. Και εμείς ε, στην αριστερά όπως είπαν πολλοί, θεωρούμε πως χρειάζεται μια ευρωπαϊκή απάντηση και ένα μηχανισμό ανακατανομή τα όσα ακούστηκαν στο πάνελ σχετικά θεωρούμε πως πρέπει πρώτα να, γίνει μια, να υπάρξει μια συμφωνία πρώτα απ' όλα αυτή η συμφωνία και μιλάμε για την ενίσχυση των εξωτερικών συνόρων. Υπάρχουν εδώ πέρα πολιτικές ομάδες που ζητάνε μια κοινή ευρωπαϊκή ακτοφυλακή. Μα ποιο το νόημα του να έχουμε κάτι τέτοιο αν δεν έχουμε ένα σύστημα διαχείρισης των ανθρώπων που φτάνουν. Αυτό πρέπει να λύσουμε και μετά να δούμε τα υπόλοιπα. Είναι λάθος να μπερδεύουμε την ελεγόμενη ασφάλεια με τα εξωτερικά σύνορα και τις λύσεις που πρέπει να βρούμε στο ζήτημα των προσφύγων. Ένας μηχανισμός λοιπόν, όπως είπαμε, κατανομής και μεγαλύτερη ευρωπαϊκή ευθύνη. Αυτό πρέπει να ζητήσουμε. Και γρήγορα κιόλας. Αντί να ασχολούμαστε με τα εξωτερικά σύνορα. Εμείς λέμε όχι στα έξυπνα σύνορα, στη Frontex, όχι στη στρατιωτική παρέμβαση μέχρι να ε, αποκτήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση μεγαλύτερη ευθύνη για την ε, κατάσταση με τους πρόσφυγες. Και βλέπω εδώ πέρα φιλμάκι πως αυτό ζητάει ο κόσμος. Ε, το ερώτημα ήταν εάν θεωρείτε ότι τα κράτη-μέλη θα πρέπει να εμπλακούν στην, ε, στο σύστημα αυτό κατανομής και η απάντηση είναι ναι, πως χρειαζόμαστε μια πολιτική προσφύγων ε, για την οποία θα μπορούμε να είμαστε περήφανοι, έτσι ώστε όταν μας ρωτάνε στο μέλλον τι κάνατε όταν γινόταν ε, πόλεμος, να μπορούμε να απαντήσουμε ότι ανοίξαμε τα σύνορά μας και καλωσορίσαμε τον κόσμο. Σας ευχαριστώ. Τον λόγο έχει η κυρία Λάουρα Φεράρα από το κίνημα των πέντε αστέρων. Πέντε λεπτά. Σα ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα σε όλου. Εγώ θα χρησιμοποιήσω τη διερμηνία και θα μιλήσω στη γλώσσα μου, τα Ιταλικά. Σήμερα μιλάμε για ένα θέμα εξαιρετικά ευαίσθητο, ένα θέμα που μάλιστα έχει συζητηθεί εδώ εις βάθος στο Ευρωκοινοβούλιο και όχι μόνο στο Ευρωκοινοβούλιο αλλά σε όλη την Ευρώπη. Πρόκειται για μια μεγάλη πρόκληση που αντιμετωπίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση και είναι ένα θέμα για το οποίο μιλάμε ως να είναι πρόβλημα και ως να είναι κατεπίγουσα ε, ανάγκη. Κάτι το οποίο εγώ υπογραμμίζω πάντα όταν μιλώ για μεταναστευτικές ροές ε, είναι το γεγονός ότι ανέκαθεν υπήρχαν από τότε που έχει είχε δημιουργηθεί ο κόσμος, σε μεταναστευτικέ ροές υπήρχαν ανάμεσα σε όλα τα κράτη-μέλη και εκτός των κρατών μελών. Τώρα, όταν μιλάμε για πρόβλημα ή για επίγουσα ανάγκη, είναι επειδή μέχρι σήμερα δεν έχουμε καταφέρει, δεν είχαμε τη δυνατότητα ή καλύτερα δεν είχαμε κατά τη γνώμη την πολιτική βούληση να βρούμε λύση, να βρούμε έναν τρόπο διαχείρισης ε, ε, των μεταναστευτικών ροών. Το να μιλάμε λοιπόν ε, για την μετανάστευση σαν να είναι επίγουσα ανάγκη μόνο είναι επικίνδυνο. Είναι επικίνδυνο γιατί μπορεί να μας οδηγήσει να λάβουμε αποφάσει βιαστικά, ε, να θέλουμε να καθησυχάσουμε άμεσα τους πολίτες μας. Αυτό σημαίνει ότι λαμβάνουμε αποφάσεις προσωρινού τύπου που μετά μπορεί να αποκτήσουν μόνιμο χαρακτήρα. Αποφάσεις όμως οι οποίες μπορεί να ληφθούν ε, και να είναι δεσμευτικέ ή περιοριστικές για τα θεμελιώδη δικαιώματα. Και έπειτα επειδή δεν είναι η σωστή λύση. Τα μέτρα τα οποία λαμβάνονται σε επίγουσες καταστάσεις τείνουν να απαντούν όχι με μια γενική ολοκληρωμένη προσέγγιση όπως προσπαθεί να το κάνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με τις εκθέσεις που είναι υποσύζητηση, αλλά προσπαθούν να δώσουν μια λύση αντιμετωπίζοντα μόνο το άμεσο πρόβλημα και υπό μια συγκεκριμένη μόνο πτυχή. Ιδιαίτερα μέχρι σήμερα αυτό το οποίο πολύ συσχετίζεται με την μετανάστευση είναι το η της ασφάλειας. Μεγάλη σχέση ανάμεσα στην ασφάλεια και στην μετανάστευση γίνεται. Ε, ε καταρχήν θα έπρεπε κατά τη γνώμη μου να λειτουργήσουμε προληπτικά για να λυθεί αυτή η σύνδεση, αυτή η συσχέτιση ανάμεσα στη μετανάστευση και την ασφάλεια είναι η ενημέρωση. Γιατί φοβάται κανείς αυτό που δεν γνωρίζει. Φοβάται όταν δεν γνωρίζει και με χαρά διάβασα ότι πολλοί, οι περισσότεροι μάλιστα από τα κράτη-μέλη έχουν απαντήσει λέγοντας ότι θέλουν μεγαλύτερη ευρωπαϊκή ολοκλήρωση και αυτό το θεωρούν ως προστιθέμενη αξία, πολιτιστική ανταλλαγή. Αυτό θα έπρεπε να είναι οι μεταναστευτικές ροές. Μια ανταλλαγή πολιτισμών, αρχών, παραδόσεων που εμπλουτίζουν η μία την άλλη, αλλά στη βάση η προϋπόθεση είναι η γνώση και η ενημέρωση, σωστή ενημέρωση. Επιπλέον, μιλάμε πολύ για συνεργασία και για αλληλεγγύη. Ε, πολλά, πολύ μεγάλα λόγια έχουμε να ακουστεί από τα κρατημέλη και από τη χώρα μου, την Ιταλία, αλλά και από την Ελλάδα. Χώρες ε, οι οποίες ε, έχουν αναλάβει τη μεγαλύτερη ε, υποχρέωση, έχουν το βάρος των, της μετανάστευσης και των προσφύγων. Μάλιστα προσωρινό μέτρο για 160.000 πρόσφυγες που υποτίθεται θα, θα επαναγκατασταθούν, αλλά μόλις 160 άνθρωποι έχουν λάβει τις σχετικές αποφάσεις και υπάρχει μεγάλη σύγχυση για τα όσα ισχύουν. Γιατί δεν λειτουργεί αυτός ο μηχανισμός, γιατί βασίζεται στον εθελοντισμό. Είναι ένα εθελοντικό μηχανισμό και εξαρτάται από τη διακριτική σχέδια των κρατών μελών. Πολλά από τα κρατή-μέλη δεν ενδιαφέρονται να υποδεχτούν μετανάστε και αυτό προκαλεί ρήξη και προβλήματα στην πράξη, στην, στην επανεγκατάσταση των μεταναστών ή, εν πάση περιπτώσει, την κατανομή των ευθυνών ανάμεσα σε όλα τα κράτη-μέλη. Και αυτή είναι και η αντίφαση που προκύπτει και για την οποία θα μπορούσαμε να μιλήσουμε αργότερα ανάμεσα σε όσου δεν θέλουν τι υποχρεωτικέ προσωστώσει γιατί θεωρεί, ο, θεωρούν ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει το δικαίωμα και δεν μπορεί να επιβάλλει τίποτα στα κράτη-μέλη και ότι θα πρέπει να γίνει σεβαστή η αρχή τη επικουρικότητα και από την άλλη πλευρά αρνείται να δεχτεί ε, μετανάστες και άρα να βοηθήσει τα κράτη-μέλη που δέχονται το μεγαλύτερο βάρος. Ε, αυτή την αντίφαση, την αδράνεια, την αδράνεια, την έλλειψη πολιτικής βούλησης μέχρι στιγμής βασίζεται η διαχείριση των μεταναστευτικών ρόλων. Κατά τη γνώμη μου, η απάντηση που μέχρι σήμερα έχει δώσει ως 28 κράτη-μέλη είναι εξαιρετικά ανεπαρκής. Ανεπαρκής. Θα έπρεπε να γίνουν πολύ περισσότερα, να ενεργήσουμε ως μία μόνο Ευρωπαϊκή Επικράτεια και όχι ως 28 κράτη-μέλη, που ο καθένας κοιτά το αυστηρά εθνικό του συμφέρον, προσπαθεί να συζητήσει, αλλά τελικά δεν ακούει ο ένας τον άλλον. Και άρα λοιπόν τα αποτελέσματα είναι αυτά που δυστυχώς ε, βλέπουμε καθημερινά. Ευχαριστώ. ευχαριστώ και τώρα συνεχίζω. Ναι. Συνεχίζουμε. με αλφαβητική σειρά και ζητούμε συγγνώμη από την κυρία Βόζεμερκ Βιονίδη που έχει δύο επίθετα αλλά αρχίζουν με βίλα λατινικό και τα δύο και είναι τελευταία στην αλφαβητική σειρά. Θα δώσουμε το λόγο στην κυρία Κιέγγε από την Ιταλία Σοσιαλιστές και Δημοκράτες να μας φύγει την κατάσταση στη Μεσόγειο. Σας ευχαριστώ. Και ευχαριστώ για την πολύ ενδιαφέρουσα αυτή συζήτηση που κατά τη γνώμη μου είναι πολύ ενδιαφέρον που γίνεται εδώ εντός του Κοινοβουλίου όπου εργαζόμαστε για αυτά τα ε, θέματα. Το βίντεο ήταν πολύ ενδιαφέρον. Καταρχήν θα ήθελα να υπογραμμίσω ορισμένα σημεία <clears throat> και για αυτό το φόβο που έχουν οι νέοι που μετά την ανεργία σε δεύτερη θέση έρχεται ο φόβος των μεταναστών. Για πολλούς και διάφορους λόγους, σε πολλούς και διάφορους λόγους οφείλονται όλα αυτά. Καταρχήν ε, είναι πολιτικής φύσης. Δηλαδή, οι πολιτικές πώς ασκούνται, πώς εφαρμόζονται και έπειτα στρέβλωση της ενημέρωσης. Και εδώ ακριβώς που είμαστε μέσα, ανάμεσα σε δημοσιογράφου, αυτό πρέπει να υπογραμμιστεί. Πολιτική φύση Δηλαδή, πώς εφαρμόζονται οι διάφορες πολιτικές στα διάφορα κράτη-μέλη και Υπάρχει ένα κοινό νήμα, η λογική της επίγουσας ανάγκης. Όταν όλες μας τις, τις πολιτικές τις βασίζουμε στη λογική της κατεπίγουσας ανάγκης, είναι λες και θεωρούμε το μεταναστευτικό φαινόμενο ένα φυσικό φαινόμενο, καιρικό φαινόμενο. Δηλαδή, αν κανείς δεν μπορεί να καταλάβει ότι πρόκειται για μια διάκοπτη ροή, η οποία στην ουσία σε κάποιες στιγμές ε, ε, παρουσιάζει περίοδους εχμής, και, και αντίστοιχα ύφεση ε, θα πρέπει να, να καταλάβουμε ότι πρόκειται για μια τέτοια μόνιμη μεταναστευτική ροή, ώστε και οι πολιτικές μας να το δεχτούν και να προσαρμοστούν σε αυτό. Να αντιστρέψουμε λοιπόν την πορεία και τελικά να εφαρμόσουμε όλες τις πολιτικές και τα μέσα που έχουμε στη διάθεσή μας με τον καλύτερο δυνατό συνδυασμό. Εσωτερική πολιτική και εξωτερική πολιτική να συνδυαστούν, να δουλέψουμε σε στρατηγικές μέσω μάκρο και βράχη πρόθεσμες και αυτό είναι και στη βάση βάση της εργασίας που κάνουμε. Εγώ είμαι συνεισηγήτρια για αυτό το θέμα, την έκθεση πρωτοβουλίας που ασχολείται με την κατάσταση στη Μεσόγειο και την ανάγκη μιας σφαιρικής ε, προσέγγισης στο μεταναστευτικό φαινόμενο. Αλλά δεν περιοριζόμαστε πλέον μόνο στη Μεσόγειο γιατί πρέπει να διευρύνουμε τη ματιά μας προς τα Βαλκάνια. Το μεταναστευτικό φαινόμενο λοιπόν είναι διάστατο και διακρατικό. Είναι ιστορικής ε, σημασίας και γι' αυτό το λόγο θα πρέπει να το αντιμετωπίσουμε όχι με συνθήματα όπως κάνουν οι λαϊκιστές και εδώ θα μιλήσω για την άκρα δεξιά γιατί στην ουσία το δικό τους λάβαρο είναι να ενεργούν ακριβώς με συνθήματα τα οποία δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Σύντομα συνθήματα, ε, σαν είναι σαν να μιλάμε κοφτά, με λίγα λόγια. Δεν δίνουμε τη σωστή εικόνα, ούτε τη σωστή διάσταση του προβλήματος και του φαινομένου Δεύτερο σημείο που θέλω να υπογραμμίσω, γιατί ακριβώς βρίσκομαι μπροστά σε δημοσιογράφους, είναι το σημείο ότι δίνεται στρεβλωμένη η πραγματικότητα. Δεν εξηγείται αρκετά καλά τι είναι το μεταναστευτικό αυτό φαινόμενο. Όταν λοιπόν η επικοινωνία γίνεται με λάθος τρόπος, μπορεί να προκαλέσει ακριβώς αντίθετο αποτέλεσμα, δηλαδή να αυξήσει τους φόβους, να αυξήσει την συνεννοησία για το τι συμβαίνει. Ε, όταν κάποιος λέει εισβολή, ε, αλλά όταν δεις τα νούμερα ε, δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Μπορεί λοιπόν να δημιουργηθούν αρνητικές στάσεις αλλά και η απόρριψη των όσων φτάνουν στην κάθε χώρα. Πιστεύω πως έχουμε την υποχρέωση η πολιτική, αλλά και όσοι είμαστε μέσα στην επικοινωνία να δίνουμε σωστά τα στοιχεία αλλά κυρίως να συμβάλλουμε θα να γίνει καλύτερα κατανοητό σε όσους δεν έχουν ποτέ επαφή, δεν είχαν ποτέ σχέση με το φαινόμενο της μετανάστευσης να καταλάβουν γιατί πράγμα μιλάμε. Σύμφωνα με τα στοιχεία της UNHCR, της ΥΠΑ της Αρμοστίας, σε ολόκληρο τον κόσμο υπάρχουν 60 εκατομμύρια πρόσφυγες και εσωτερικά εκτοπισμένοι. Το 86% των προσφύγων βρίσκουν ε, καταφύγιο στις διπλανές τους χώρες, στις ε, γειτονικές χώρες. Ήδη μιλάμε για τα εξωτερικά μας σύνορα. Θα πρέπει να καταλάβουμε κάπως τις διαστάσεις αυτού του φαινομένου για να μπορέσουμε να δώσουμε έτσι, να συμβάλλουμε στην επεξεργασία των πολιτικών. Μιλάμε για χώρες όπως το Πακιστάν, την Αιθιοπία, το Σουδάν, την Κένια, που από μόνες, σας, τους έχουν δώσει ε, άσυλο σε 2.800.000 πρόσφυγες, δηλαδή αντίστοιχο με το 24% του παγκοσμίου προσφυγικού πληθυσμού, για να μην μιλήσουμε για την Τουρκία, τη Συρία ή το Λίβανο, ενώ στην Ευρώπη φτάνουν κάτω από το 10% των των άσυλων. Μπορούμε λοιπόν να αλλάξουμε τη στάση μας, γιατί όταν λέμε ότι αντιμετωπίζουμε μια κρίση, ναι, αλήθεια είναι κρίση όταν από τη μια πλευρά βλέπουμε μια ξαφνική άφηξη μεταναστών. Θα πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι η πραγματική κρίση είναι το πολιτικό αδιέξοδο στο οποίο βρίσκεται η Ευρώπη και η μοιοπία των κρατών μελών. Γιατί πολλές φορές όταν μιλάμε βάζουμε όλους το ίδιο καλάθι, το Κοινοβούλιο, την Κομισιόν και το Συμβούλιο. Εδώ πρέπει να υπογραμμίσουμε πως το Ευρωκοινοβούλιο κάνει δουλειά με προτάσεις πολύ συγκεκριμένες ενώ χτυπάμε μπροστά, συγκρουόμαστε με το τείχο των εγωισμών των κρατών μελών και πρέπει αυτό να το εξηγήσουμε. Μειοπικά τα κράτη-μέλη που πεισματικά δεν θέλουν να εκπονήσουν μια μακροπρόθεσμη στρατηγική κοινή στρατηγική και από αυτού πρέπει να δουλέψουμε περισσότερο. Εμείς είμαστε βουλευτές, αντιπροσωπεύουμε, είμαστε άμεσα εκλεγμένοι από τους λαούς και θέλουμε τη φωνή των λαών να μεταφέρουμε εδώ και έχουμε την υποχρέωση να καταφέρουμε να υποβάλουμε προτάσεις που να αντιπροσωπεύουν ακριβώς τους πληθυσμούς που μας έχουν εκλέξει. Όσον αφορά το σύστημα των ποσοστώσεων, εγώ προσωπικά είμαι υπέρ ενός μόνιμου μηχανισμού αλληλεγγύης και κατανομή των ευθυνών σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Δηλαδή ε, είμαι υπέρ ενό νομοθετικού νομοσχεδίου Προς αυτό θα πρέπει να προχωρήσουμε, αλλά χρειάζονται και μέσα που θα κινητοποιήσουν προς την αντιμετώπιση του συστήματος και άρα ένα σύστημα ε, των ποσοστώσεων. Θα ήθελα επίση να επιμείνω στις νόμιμε όδου μετανάστευση. Ανάμεσα στις λύσεις που προτείνονται θα πρέπει να επιμείνουμε στο γεγονό ότι πρέπει να δημιουργηθούν νόμιμοι δρόμοι, γιατί και αυτό θα ήταν μια λύση ώστε να ξεφύγουν από τα χέρια των διακινητών οι μετανάστες που δεν βρίσκουν άλλη λύση από το να αφήσουν τη ζωή του στα χέρια των λάθο ανθρώπων. Ευχαριστώ. Uh, maybe, maybe I didn't say δεν το είπα ε, προηγουμένως, θα δώσουμε το λόγο στην κυρία Βόζεμπερκ που είναι από την Ελλάδα, από το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, Χριστιανοδημοκράτες και αντιπρόεδρος της Ομάδας Εργασίας ε, Νομικών Υποθέσεων και Εσωτερικών. Θα μου επιτρέψετε να μιλήσω στην μητρική μου, παρακαλώ. Ε, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, Σήμερα που συζητούμε είμαστε στη σκιά ενός άλλου τραγικού γεγονότος. Σήμερα το πρωί περισυνελέγησαν 12 πτώματα πάλι στο Φαρμακονήσι, στα Δωδεκάνησα, στην πατρίδα μου, εκ των οποίων έξι ήταν μωρά, 4 ε, άνδρες και δύο γυναίκες. Αυτό είναι ένα φαινόμενο που καθημερινά εμφανίζεται. Ξέρετε ότι το Αιγαίο και η Μεσόγειος ευρύτερα έχει χαρακτηριστεί σαν ένα απέραντο νεκροταφείο εδώ και ένα χρόνο θα διαρωτηθούμε η μετανάστευση και το προσφυγικό, δεν κάνω διάκριση, αλλά είναι ένα ενιαίο πρόβλημα. Χτύπησε την πόρτα της Ευρώπης σήμερα. Όχι βέβαια. Απλώς οξύνθηκε τον τελευταίο χρόνο και επιτέλους η Ευρωπαϊκή Ένωση κατάλαβε ότι δεν είναι ένα πρόβλημα που αφορά στο Νότο επειδή στο Νότο παρουσιάζονταν τα αυξημένα μεταναστευτικά ρεύματα αλλά όταν οι άνθρωποι αυτοί απελπισμένοι χτύπησαν την πόρτα της κεντρικής και της βόρειας Ευρώπης η Ευρώπη αντελήφθη ότι χρειάζεται μια ολιστική, γενική, ευρωπαϊκή πολιτική σε μεταναστευτική κατεύθυνση αλλά πάντοτε με, με ανθρωπιστικό χαρακτήρα. Αυτό τι σημαίνει πολύ απλά, ότι ευνηδιάστηκε η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αν δεν ευνηδιάστηκε, τότε ολιγόρησε. Όταν ευνηδιάστηκε όμω, ποιε αποφάσει πήρε. Οφείλω να πω ότι λήφθησαν κάποιε σημαντικέ αποφάσει. Είναι όμω δεσμευτικού χαρακτήρα. Έχουν λύσει το πρόβλημα ή απλώ το διαχειρίζονται πάνω στην οξύτητά του. Θα σα πω λοιπόν πολύ απλά ότι οι αποφάσει τι οποίε πήραμε για τη μετεγκατάσταση στα κράτη-μέλη την αναδιανομή με βάση συγκεκριμένα αντικειμενικά κριτήρια που αφορούν είτε τις οικονομικές συνθήκες, είτε τις θέσεις εργασίας, είτε τις ανάγκες κάθε κράτους μέλους, είναι μια σωστή απόφαση υπό την προϋπόθεση ότι θα βρει ανταπόκριση αφενός μεν στην αλληλεγγύη, μέχρι στιγμής δεν το έχουμε δει από όλα τα κράτη-μέλη, και αφετέρου να προωθηθεί σε ένα μόνιμο δεσμευτικό μηχανισμό, δηλαδή να έχει το χαρακτήρα οδηγίας που θα έχει μια δεσμευτικότητα για τα κράτη-μέλη. Μέχρι στιγμής, όπως είπαμε, επαφίεται στην αλληλεγγύη, η οποία ολιστικά και συνολικά δεν λειτουργεί. Το δεύτερο μέτρο της επανεγκατάστασης, δηλαδή του resettlement από τι από τις τρίτες χώρες που θεωρούνται ασφαλείς και όμως καλύπτουν κενά στην Ευρωπαϊκή Ένωση με βάση τα κριτήρια που θα έχουν βρεθεί, δηλαδή τις ανάγκες, τα εργασίες και το εξειδικευμένο δυναμικό και αυτή η απόφαση είναι σωστή υπό την προϋπόθεση ότι και αυτή θα μπορεί να έχει μια δεσμευτικότητα και μια οριστική εφαρμογή όχι ως διαχείριση αλλά ως αντιμετώπιση του προβλήματος. Αυτές οι αποφάσεις όπως ξέρετε ελήφθησαν μόλις πρόσφατα. Δηλαδή πάντοτε μιλάμε για το τελευταίο οκτάμινο-δεκάμινο. Πώς μπορεί όμως, ε, κυρίες και κύριοι, να ρυθμιστεί το θέμα της ε, μετανάστευσης και ιδιαίτερα το προσφυγικό. Είναι ένα θέμα που ανέκυψε στην οξύτητά του τώρα, αλλά ξέρουμε ότι τα φαινόμενα που το δημιούργησαν, με άλλα λόγια και ο πόλεμος μένεται 4,5 χρόνια και γενικά η μετανάστευση που αναφέρεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να έχει τώρα μια οξύτητα, αλλά έχει και μια διαχρονικότητα. Και το πρόβλημα δυστυχώ ήρθε για να μείνει. Καλείται λοιπόν η Ευρωπαϊκή Ένωση να διερωτηθεί όλες οι πολιτικές ομάδες, όλες οι πολιτικές τάσεις, όλοι οι προβληματισμοί, όλες οι ιδεολειψίες ή οι ιδεολογίες ή οι αγγυλώσεις που υπάρχουν ενδεχομένως, δεν κατηγορώ κανένα, βάζω προβληματισμούς, μπορούν να συμφωνήσουν ότι χρειάζεται μια ενιαία ευρωπαϊκή πολιτική. Και πώς θα το συμφωνήσουν αν οι πολιτικές ομάδες δεν το επιτρέψουν. Έχει ανοίξει ένας ευρύς διάλογος, θέλω να πιστεύω. Μεθαύριο, το μεθαύριο το λέω σχηματικά αλλά είναι σύντομα, θα ψηφιστεί η η οδηγία που έχει ανάγκη η Ευρωπαϊκή Ένωση για το PNR, για τα δεδομένα των επιβατών. Μέχρι στιγμής έχουν ληφθεί αποφάσεις. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υπάρχει η πλειοψηφία. Αλλά αυτό για να γίνει οδηγία χρειάζονται ακόμη βήματα. Το λέω γιατί στο πολύ ενδιαφέρον φιλμάκι που είδαμε με τα στατιστικά βλέπουμε ότι το 72% των Ευρωπαίων πολιτών θεωρούν ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει μεγάλη σημασία από τότε που βάσει της ε, συνθήκης της Λισαβόνας συνομοθετεί. Επομένως, εκεί όπου χρειάζεται να συμβάλλει σε μια νομοθεσία, θα πρέπει να συνδράμουν όλες οι πολιτικές ομάδες και να συνδράμει όλη η Ευρωπαϊκή Ένωση ανάλογα με τις νοοτροπίες των κρατών μελών και με οποιαδήποτε ιστορικές αναδρομές μπορούν να εξηγηθούν, να καταλάβουν ότι είναι ένα κοινό μας πρόβλημα. Αυτή τη στιγμή αντιλαμβάνεστε, σας μιλώ ως Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα και δεν μιλώ απλώς ως Ελληνίδα, διότι αν μιλούσα ως Ελληνίδα θα σας έλεγα ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση όφιλε να μην είναι τόσο ευέλικτη στον στρατηγικό εταίρο που ονομάζεται Τουρκία όταν γνωρίζουμε ότι τα τεράστια μεταναστευτικά ρεύματα πια έρχονται στα παράλια, από τα παράλια της Τουρκίας στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και μέσω της Ελλάδος να καλούνται να διανεμηθούν οι άνθρωποι αυτοί και δεν αιτιώμε ενδεχομένως κάποια λάθη της όποιας ε, Ελλάδος, της όποιας χώρας που είναι η χώρα μου, αλλά αιτιώμε την αναγκαιότητα να υπάρχει ίση αντιμετώπιση στα κράτη-μέλη που έχουν την οξύτητα του προβλήματος, ούτως ώστε ολιστικά και πανευρωπαϊκά να ρυθμιστεί. Τα επόμενα βήματα που πρέπει να κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση και στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα έχουμε τέτοιες αποφάσεις, είναι εντός του, του Μαρτίου του μέχρι το Μάρτιο του 2016 να επανεξεταστεί το Δουβλίνο 2-3, το όποιο Δουβλίνο ισχύει αυτή τη στιγμή αφού τα πραγματικά γεγονότα το έχουν ξεπεράσει, να οριστεί πλέον, να καθοριστεί και να προσδιοριστεί η επανεγκατάσταση από τις τρίτες χώρες και βεβαίως μια αναθεώρηση συνολικής στρατηγικής υπό την προϋπόθεση ότι αντιλαμβανόμαστε όλη την αναγκαιότητα να φυλάσσουμε κυρίες και κύριοι τα εξωτερικά μας σύνορα. Και όσοι πιστεύουν ότι ενδεχομένως το PNR όταν οριστικοποιηθεί ή οποιασδήποτε ε, ε, αποφάσεις λαμβάνονται για τη θωράκιση της ασφάλειας των πολιτών τυχόν γιατί ακούμε τέτοιες φωνές θέτουν εν κινδύνο τα θεμελιώδη δικαιώματα, θα σας πω με το χέρι στην καρδιά και με πεποίθηση από τις νομικές μου γνώσεις ότι η ασφάλεια του πολίτη, το ξέρουμε όλοι, αντίθετα θωρακίζει τα θεμελιώδη δικαιώματα και προάγει την ελευθερία του πολίτη, διότι ο ανασφαλής πολίτης είναι ο φοβικός πολίτης, εκείνος που δεν μπορεί την επόμενη στιγμή να είναι ελεύθερος. Οπωσδήποτε δεν θα συνδυάσουμε ποτέ τη μετανάστευση με την τρομοκρατία άμεσα, αλλά δεν θα παρα παραβλέψουμε και το γεγονός ότι μέσα από τα μεταναστευτικά ρεύματα παρισφρέουν άτομα τέτοια τα οποία έχουν τις ιδιότητες αυτές διότι αντιλαμβανόμαστε ότι και το πρόσφατο χτύπημα στην Γαλλία χαρακτήρισε Ευρωπαίους πολίτες. Πολίτες οι οποίοι είχαν ευρωπαϊκά διαπατήρια και άρα είχαν εκπαιδευτεί με έναν τρόπο ακριβώς για το σκοπό αυτό. Αυτό σημαίνει ότι είμαστε, δεν θα αλλάξουμε ποτέ ως Ευρώπη την πολιτική των ανοιχτών συνόρων, της ελεύθερης διακίνησης των ιδεών και των ανθρώπων υπό την προϋπόθεση ότι τα σύνορά μας θα είναι ελεγχόμενα από εμά τους ίδιους με κανόνες που θα εξασφαλίζουν την αλληλεγγύη των Ευρωπαίων πολιτών και την πολιτική βούληση να υπάρχει μια ολιστική συνεκτική πολιτική που θα καλύπτει την Ευρώπη και θα θωρακίζει την ελευθερία της ενδυναμώνοντας και το ρόλο της και τελειώνοντας να πω ότι γι' αυτό απαιτείται τόσο συνεργασία με τις χώρες προέλευσης των ανθρώπων αυτών όσο και άμεση συνεργασία με τις χώρες διέλευσης, ιδιαίτερα όταν καλούνται να έχουν το ρόλο του στρατηγικού εταίρου. Σας ευχαριστώ πολύ. Έχω μια ερώτηση για την Ευρώπη. Μήπως να σταματήσουμε προς το καλό της Ευρώπης να χρησιμοποιούμε τον όρο Γιατί γιατί έρχεσαι στις Βρυξέλλες και αρχίζει και ολιστική προσέγγιση ακόμα και όταν πας στο μπακάλι. Ας πούμε, να το πούμε κάπως αλλιώς, δεν το λέω για σας. Όλοι χρησιμοποιούν αυτή την ολιστική... Ε, ό,τι δεξιά και αριστερά ακούς θέλουμε μια ολιστική προσέγγιση. μα, σας εξήγησα, λέει η κυρία τι εννοώ. Ε, εντάξει, λοιπόν, 25 λεπτά ερωτήσεις. Έχετε το λόγο. Εσείς παρακαλώ. Παρακαλώ με μικρόφωνο. Θα ήθελα... Ε, από το Micron Report είμαι, Μάρτιν ε, Γκάλ. Θέλω να κάνω μια ερώτηση σε όλο το πάνελ για τη συμφωνία με την Τουρκία. Ε, είπε η κυρία Βόζεμπεργκ ε, τι συμβαίνει σήμερα και στο φαρμακονίσι το δράμα που είχαμε. Εγώ μόλις επέστρεψα από την Τουρκία και έχει καταρρεύσει η κατάσταση στην Τουρκία. Από το Ποντρούμ τους πηγαίνουν ε, σε διαδρομές που είναι πιο μακριές και πιο επικίνδυνες. Και θα ήθελα να μας απαντήσει το πάνελ ε, για τη συμφωνία που επετεύχθη σε δύο επίπεδα. Πρώτον, από πλευράς οικονομικής και την τουρκική πρόπτικη, αν δούμε τους αριθμούς, πριν από πέντε χρόνια υπολογίστηκε ότι η Τουρκία θα πρέπει ε, να δαπανά 23.000 ευρώ αναπρόσφυγα για την περίθαλψή του, την κάλυψή του, την ασφαλιστική κτλ. Εάν χρησιμοποιηθεί αυτό το στοιχείο τα 3 δισεκατομμύρια, ε, ε, καταλαβαίνετε σε τι αντιστοιχούν. Ε, φτάνουν για 130.000 ενώ είναι 2 και 2,5 εκατομμύρια οι πρόσφυγες. Το δεύτερο, σε ό,τι αφορά την Τουρκία αν είναι αξιόπιστος εταίρος. Αυτή τη στιγμή ουδής, ουδής, ούτε Σύρος, ούτε Αφγανός, ούτε Ιρακινός μπορεί να πάρει το καθεστώς πρόσφυγα. Αυτό που ζητούν οι άνθρωποι στην Τουρκία. Είναι ένα μέλλον, μια προοπτική. παρόλο που ανταποκρίνονται στα κριτήρια της Σύμβασης της Γενέβης, δεν υπάρχει δυνατότητα απονομής του καθεστώτος πρόσφυγα. Την εθνικότητά σας δεν άκουσα. Είστε Τούρκος. Όχι, όχι, Μαλτέζος είμαι, αλλά ε, μόλις επιστρέφω από την ε, Τουρκία. Ε, για τα οικονομικά λοιπόν και για τους πρόσφυγες τι γίνεται με τη συμφωνία. Ποιος θέλει να απαντήσει, ποια κυρία μάλλον. Κοιτάξτε, επειδή μπορεί να έχουμε διαφορετικές απόψεις, εμείς στην ομάδα της αριστεράς επικρίνουμε αυτή τη συμφωνία γιατί την θεωρούμε ένα στοιχείο με το οποίο η Ευρωπαϊκή Ένωση προσπαθεί να αναθέσει σε άλλους τα σύνορά τους, σε τρίτες χώρες δηλαδή, να είναι υπεύθυνε για να ανασχέσουν αυτή τη ροή. Ε, το λέει όμα θέλει οι αφρικανικές χώρες ο κύριος Τούσκ να σταματήσουν ε, οι Αφρικανοί να έρχονται στα ευρωπαϊκά σύνορα και το ίδιο με την Τουρκία. και νομίζω πως ε, στο ευρωπαϊκό ε, επίπεδο βλέπουμε πως η Τουρκία δεν σέβεται την ελευθερία των ε, ΜΜΕ, δεν τα πάει καλά στα ανθρώπινα δικαιώματα, μειωματικά δικαιώματα. Και κάνουμε τα στραβά μάτια εμείς για την καταστολή της κουρδικής μειονότητας. και ακόμα αφήσαμε, επιτρέψαμε και στον Ερντογάν να αυξήσει την καταστολή αυτή μέσα και έξω από την ε, Τουρκία. Ανησυχούμε για το τι γίνεται. Η Human Rights Watch λέει πως ε, γίνονται, κάνει αποθήσεις ε, σύρων στα σύνορα που προσπαθούν δηλαδή να μπουν στην Τουρκία και τους αποθούν και τους φυλακίζουν και είναι απαράδεκτη κατάσταση Οπότε η συμφωνία αυτή είναι ηθικά και πολιτικά και πρακτικά δεν θα κάνει αυτό το οποίο θέλει ο Ντόναλντ Τούσκο και είναι ντροπή για τους Ευρωπαίους ηγέτες. Ε, Από τη σειρά μου να απαντήσω πέραν του γεγονότος ότι έκανα μια αναφορά ε, στο θέμα αυτό. Η Ευρωπαϊκή Ένωση οπωσδήποτε θεωρεί στρατηγικό εταίρο την Τουρκία, αλλά σίγουρα και στην πολιτική μας ομάδα το έχουμε επισημάνει, πρέπει να ασκηθεί περισσότερη πίεση, γιατί ξέρουμε ότι η Τουρκία, ε, αν μη τι άλλο, ούσα σε προενταξιακή ε, πορεία, δεν τηρεί τις συμφωνίες επανιστοχής, ζητάει, ε, προβάλλει συνέχεια αιτήματα, όπως και οικονομικά, έχει ήδη εγκριθεί να πάρει 3 δισεκατομμύρια επιπρόσθετα για το θέμα αυτό και ζητάει ελάφρυνση της βίζας για τους πολίτες. Λοιπόν, θα πρέπει να αντιληφθεί οποιοδήποτε βρίσκεται σε αυτή την ε, προενταξική πορεία ότι αν δεν τηρούνται οι προϋποθέσεις της Κοπενχάγης θα πρέπει να συμμορφωθεί, υπάρχουν ίσοι όροι όταν υπάρχουν συναλλαγές αυτού του επίπεδου. Ευχαριστώ πολύ.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 προβληματισμένοι και από οικονομικές άποψεις αλλά και όσον αφορά τα ανθρωπιστικά ζητήματα. Τους υποσχεθήκαμε τρία δις για τους προσφυγικούς καταβλισμούς όπου προστίθεται τα κονδύλια τα προενταξιακά και από το προηγούμενο πρόγραμμα και από το καινούριο φτάνουμε σχεδόν σε 9 δις ευρώ που δίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση σε μια χώρα που δεν είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση ακόμα. Όταν όσον αφορά την αξιοπιστία και τα ανθρώπινα δικαιώματα θα είχαμε πολλά να πούμε. Εγώ πραγματικά έμεινα με ανοιχτό το στόμα όταν ο Γιούνκερ στην Ολομέλη μα είπε ότι η Τουρκία είναι μια σίγουρη χώρα, αξιόπιστη και ότι θα μπει στον κατάλογο των ασφαλών χωρών. Παρά τα τόσα που φτάνουν τα νέα σε σχέση με την παραβίαση των θεμελιωδών ανθρωπιστικών, ανθρωπινών δικαιωμάτων, ε, διώξεις ε, κατά των Κούρδων, αλλά και άλλων. Εγώ και η ομάδα μου και η αντιπροσωπεία του κινήματος 5 αστέρων ε, δεν συμφωνούμε με αυτή τη συμφωνία με μια χώρα που φαίνεται να είναι και πολύ κοντά στις ε, τρομοκρατικές οργανώσεις που εμείς ε, ε, πολεμούμε. Είμαστε σε βαθιά διαφωνία μάλιστα. Γιατί Κατά τη γνώμη μα δεν είναι ο σωστός τρόπος για να αντιμετωπίσουμε τις μεταναστευτικές ροέ. Δεν είναι ο σωστός τρόπος. Ο σωστός τρόπος θα έπρεπε να είναι να αναλάβουμε τις ευθύνε των όσων κάνουμε. Να προσπαθήσουμε να ε, αντιμετωπίσουμε τις πηγές και όχι να προσπαθούμε να βουλώσουμε τρύπε, να προσπαθούμε να καλύψουμε τα προβλήματα που συχνά οι ίδιες οι ευρωπαϊκές χώρες προκαλούν. Να προσπαθούμε να τα κουκουλώνουμε και να ανύπτουμε τα σχήρας μας, δίνοντα χρήματα στου άλλου για να βρουν αυτή τη λύση. Αυτή είναι η θέση μας. Ευχαριστώ. Eh, η δική μου θέση είναι λίγο διαφορετική γιατί γνωρίζουμε ότι παρότι υπάρχουν σοβαρές αντιφιβολίες για την κατάσταση που επικρατεί στην Τουρκία, δεν μπορούμε να ξεχνάμε ότι πρέπει και να προσπαθούμε τουλάχιστον να την συμπεριλαμβάνουμε στην εξέβρεση, στην προσπάθεια εξέβρεση μια λύση. Και το λέω γιατί αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να κάνουμε πως δεν βλέπουμε ότι στην Τουρκία υπάρχουν ένα σωρό πρόσφυγε, ένα σωρό κόσμο, ε, του οποίου πρέπει να βοηθήσουμε, να του υποδεχτούμε, αν και εξακολουθούμε να καταγγέλουμε. Η ομάδα μας δηλαδή έχει τη θέση ότι αυτή η συμφωνία δεν αρκεί, ότι θα πρέπει να κάνουμε περισσότερα, αλλά δεν μπορούμε πάντως να αποκλείσουμε την Τουρκία από την ε, αναζήτηση μιας απάντησης και μιας λύσης. Πρέπει να μπούμε στη βαθιά αίτια των όσων προκαλούν τη μετακίνηση των ανθρώπων αυτών, αλλά στη γενική και σφαιρική στρατηγική και στην εξέβρεση λύσης πρέπει να υπάρχει και η Τουρκία. Ναι, να βρεθεί λύση στις σειράξεις, αλλά και με την Τουρκία μαζί. Αυτό στο οποίο πρέπει να επιμείνουμε είναι η προστασία και ο σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, αλλά να ζητήσουμε από την Τουρκία και το σεβασμό των δεσμεύσεων, κυρίως από αυτέ τι βάσει. Δεν μπορούμε να την αφήσουμε όμω απ' έξω. Λοιπόν, ε, στο 7 να βάλουμε τα δυνατά μας να επιταχύνουμε λίγο. Ε, καλημέρα σας. Κάνω Λανία από το Ιταλική Εφημερίδα Μανιφέστο. Αυτά όσα είπατε με οδηγούν να υποβάλω μια ερώτηση. Από ακούμε για μια Ευρώπη πολύ αλληλέγγυη απέναντι στους μετανάστες, ενώ ταυτόχρονα ακούμε να γίνεται λόγος για την ανάγκη ενίσχυσης των εξωτερικών συνόρων της Ένωσης. Συμφωνίες με την Τουρκία αλλά και με την Αφρικανική Ένωση, με την διάσκεψη κορυφής της Μάλτας, έτσι ώστε να μας βοηθήσουν να αποφύγουμε τις αναχωρήσεις από εκεί, εκτός που είναι αντίφαση αυτό όλο. Ε, παράδοξο, είναι και υποκριτικό από πλευρά τη Ευρώπη, ε, δεν είναι. Δηλαδή, από τη μια κάνουμε ότι είμαστε αλληλέγγυοι, αλλά τελικά ο πολιτικό στόχο είναι να σταματήσουμε τι αναχωρήσει, να εμποδίσουμε του μετανάστε, άσχετα με το αν είναι πρόσφυγε ή οικονομικοί μετανάστε. Στην πραγματικότητα, ο πραγματικό στόχο είναι στο όνομα μιας ανθρωπιστικής πρωτοβουλίας να εμποδίσουμε τις αναχωρήσεις, να μείνουν εκεί που βρίσκονται. Αν και, όπως είπαμε και στην Τουρκία, με αμφισβητήσιμους τρόπους γίνονται όλα αυτά. Την ημέρα μετά τη συμφωνία με την Τουρκία συνελήφθησαν 1.300 μετανάστες από την τουρκική ακτοφυλακή. Ευχαριστώ. Ε, σε ό,τι με αφορά, εγώ θα σας πω ότι εκ διαμέτρου αντίθετη ήταν η δική μας τοποθέτηση. Αναμφίβολα δεν θέλουμε να εμποδίσουμε τους ανθρώπους αυτούς που θέλουν να βρουν ε, μια αξιοπρεπή διαβίωση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι κάτι άλλο που είπαμε. Είναι τελείως διαφορετικό να ασκείται μια πολιτική της εισρωής ανεξέλεγκτα ανθρώπων οι οποίοι άλλοι δικαιούνται να έχουν την ιδιότητα του πρόσφυγα και άλλοι είναι απλώς οικονομικοί μετανάστες και τελείως διαφορετικό να υπάρχει μια δίκαιη κατανομή στα κράτη-μέλη υπό την προϋπόθεση ότι και αυτά θα δείχνουν αλληλεγγύη ανάλογα με το οικονομικό μέγεθος του κάθε κράτους μέλους, το ακαθάριστο εθνικό προϊόν και τις θέσεις εργασίας, ούτω ώστε να μπορούμε ότι η Ευρώπη υποδέχεται ανθρώπους, αλλά έχει και τη δυνατότητα να τους παρέχει αξιοπρεπείς συνθήκες διαβίωσης. Δεν θα μπορέσει να τους στηβάζει σε κάποια μέρη, διότι δεν αδυνατεί κάτι άλλο να κάνει. Είναι τελείως διαφορετικό. Μιλήσαμε για μετεγκατάσταση και για επανεγκατάσταση. Και αναδιανομή στα κράτη-μέλη και από τα τρίτα, ε, με βάση συγκεκριμένα συγκεκριμένα κριτήρια. Αρκεί να υπάρχει αλληλεγγύη. Αυτό επικαλέστηκα τουλάχιστον εγώ. Ε. Ναι, ναι, εγώ θα ήθελα να απαντήσω. Αλληλεγγύη και έλεγχος. Ναι, είναι η μεγάλη αντίφαση που υπάρχει αυτή τη στιγμή στην Ευρωπαϊκή Ένωση και είναι και η μεγάλη υποκρισία ε, επίσης που ε, μεταφράζεται σε αυτή τη δίθεν καλοπροαίρετη θέση, ας τους βοηθήσουμε αλλά στα σπίτια τους, στη χώρα τους. Δηλαδή, ε, ναι, ναι, να τους βοηθήσουμε αλλά να μείνουν σπίτια. Πώς δεν τους δώσουμε λεφτά, δεν έχει σημασία ποιο θα τα πάρει, πώ θα χρησιμοποιηθούν, τι είδου project χρηματοδοτούνται και τι αποτελέσματα πετυχαίνουμε. Το σημαντικό είναι να πούμε ότι ναι, εμεί δίνουμε ένα δι 300 για την Αφρική, ενώ δίνουμε τρία δι στην Τουρκία γιατί που θα μα βοηθήσει για του πρόσφυγε. Και έτσι νομίζουμε ότι του βοηθάμε. Ενώ θα έπρεπε να γίνεται κάτι τελείω διαφορετικό. Το να του βοηθήσουμε στη χώρα του θα μπορούσε να ισχύει, ναι, αν και να το συμμεριζόμαστε, εάν μεταρρυθμίσουμε αν μπορέσω, μπορούσαμε να σταματήσουμε το να αισθάνονται υποχρεωμένοι να φύγουν οι άνθρωποι αυτοί. Να αλλάξουμε δηλαδή την ζωή τους εκεί. Αυτό που έλεγα πριν που αφορά στην συνέπεια ανάμεσα στο να προωθήσουμε λύσεις ενώ ταυτόχρονα εμείς προκαλούμε τα πρόβλημα. Εάν θέλουμε να τους βοηθήσουμε να μείνουν στις χώρες τους και να μην υποχρεώνονται να φύγουν, θα πρέπει να ξεκινήσουμε λέγοντας όχι στην εκμετάλλευση των φυσικών τους πόρων. Πρέπει να ξαναδούμε τις εμπορικές μας πολιτικές, τις ενεργειακές μας πολιτικές. Να λέμε όχι στην εκμετάλλευση των ανθρωπίνων πόρων τους, όχι στη βόληση των όπλων. Και να αναλάβουμε την ευθύνη με μια ισχυρή πολιτική βούληση, γιατί θα πρέπει έτσι να δούμε τα τα αίτια που υποχρεώνουν όλον αυτόν τον κόσμο να φεύγει γιατί έτσι θα μπορούσαμε πραγματικά να τους βοηθήσουμε να μείνουν σπίτια τους και να έχουν την ευκαιρία να μην αφήσουν τη χώρα τους, να ζήσουν αξιοπρεπώς στην ίδια τους τη χώρα, να προστατεύσουμε τα βασικά τους ανθρώπινα δικαιώματα και να διαχειριστούμε με πιο αποτελεσματικό και κανονικό τρόπο τις μεταναστευτικές ροές. Ωραία. Ολιστική προσέγγιση της Ευρωπαϊκής ε, Ένωσης. Έχουμε άλλα πέντε λεπτά, σύνολο οκτώ, γρήγορα. Γεια σας. Ράιν Κόλλη λέγομαι, από την Εσθονία, μικρή χώρα στη Βόρεια Ευρώπη και εργάζομαι ε, για ε, έναν τηλεοπτικό σταθμό. Θέλω να ρωτήσω κάτι για την επανεγκατάσταση και τη μετεγκατάσταση. Το πρόγραμμα ε, είναι διπλό πρόγραμμα δημοσίων σχέσεων. Πρώτο, πρέπει να πουλήσετε εντό εισαγωγικών την ιδέα ότι έρχονται μετανάστες και είναι τμήμα της κοινωνίας μας σε ανθρώπους που ζουν στα κράτη-μέλη. Αυτό είναι το πρώτο μήνυμα. Και το δεύτερο είναι που πρέπει να πουλήσετε και πάλι εντό εισαγωγικών την ιδέα ότι θα μετακατασταθούν και όλα ή θα επανακατασταθούν ήδη οι πρόσφυγες. Και α είμαστε ειλικρινεί, κάποιες χώρες της ευρωπαϊκή Ένωση είναι πολύ πιο πρόθυμε από κάποιες άλλες. Η δική μου χώρα, για παράδειγμα, είναι μικρή, είναι φτωχή, είναι μικρά τα επιδόματα, ο καιρός όχι και τόσο καλός και πολλοί άνθρωποι είναι εχθρικοί και προ του ίδιου του γειτονές τους. Ερώτηση λοιπόν, δεν θα έπρεπε να υπάρχει, θα έπρεπε να υπάρχει δυνατότητα επανεκατάστασης και μετακίνησης των μεταναστών, των προσφύγων σε χώρες που δεν θέλουν να πάνε οι άνθρωποι. Δηλαδή αναγκαστική επανεκατάσταση. Γι αυτό, μιλήσαμε για αντικειμενικά κριτήρια. Αυτό το οποίο περιγράψατε θα συμπεριλαμβάνεται στα αντικειμενικά κριτήρια. Οι ποσοστώσεις για τις οποίες μιλήσαμε δεν θα είναι, δεν θα είναι ανεξαρτήτως των αντικειμενικών κριτηρίων. Αν πράγματι η χώρα σας έχει πολύ συγκεκριμένες ανάγκες ή καθόλου ανάγκες θα ληφθεί υπόψη. Δεν πρόκειται να επιβληθούν σε ένα κράτος μέλος οι ξένοι αυτοί άνθρωποι όταν το κράτος μέλος αδυνατεί αντικειμενικά είτε για λόγου οικονομικούς είτε για άλλου λόγους να τους υποδεχτεί και να τους φιλοξενήσει. Αυτός είναι και ο στόχος του δίκαιου μέτρου αυτού. Διαφορετικά δεν θα μπορέσει να εφαρμοστεί. Eh, ναι, η ανακατανομή είναι μια πρόταση που την έχουμε προτείνει να λάβουμε υπόψη και τη βούληση του ετούντος άσυλο. Δηλαδή είναι κριτήρια τα οποία εμείς ως Κοινοβούλιο περιλάβαμε στην πρόταση, τροποποιώντας την πρόταση του Συμβουλίου και ζητήσαμε να το λάβει υπόψη. Πρέπει να λάβουμε επίσης την οικογενειακή επανένωση, δηλαδή τη δυνατότητα να μπορεί κανείς ε, να συγκεντρώσει όχι μόνο το ευθυνό αλλά και την ευρύτερη κοινότητα. Πολλές ε, δεσμεύσεις δηλαδή, πολλές ε, προβλήματα που πρέπει να ληφθούν υπόψη, πέρα από την ανακατανόμη του πληθυσμού, τη διάσταση της χώρας, είναι θέματα όλα αυτά που πρέπει να ληφθούν υπόψη όταν μιλάμε για την ανακατανομή των ετών των άσυλο σε επίπεδο των 28 χωρών. Είναι ευρέως γνωστό ότι στη Σουηδία έχει πάντα καλοκαιρία. Ε, ε, είχα πάει στα Βαλκάνια και ρώτησα κόσμο από πού είστε, από πού πηγαίνετε και μου λέγανε όλοι Σουηδία, Γερμανία, μπορεί και Βέλγιο, μπορεί και Ολλανδία, θα δείξει. Και κανείς δεν μου είπε Εστονία. Έχετε δίκιο σε αυτό που λέτε. Ε, και επίσης εξεπλάγει, κανεί δεν θα πάει στη Γαλλία από όλου αυτού. Εγώ θα λυπόμουν του Γάλλου για την εικόνα που δίνουν. Δηλαδή και εδώ χρειάζεται δουλειά να γίνει. Υπάρχει δυσκολία με το μηχανισμό αυτό, για τον αναγκαστικό πραγματικά. Και αυτό είναι ένα από τα προβλήματα για την επανεκατάσταση των 160.000 σήμερα. Πρέπει να βρούμε δηλαδή ένα τρόπο πολύ πιο ευφυή, πιο εύστοχο και να ρωτάμε και τον κόσμο που θέλουν να πάνε και πώς μπορούμε να τους βοηθήσουμε και να τους υποστηρίξουμε να αρχίσουν μια ζωή στην Ευρώπη. Ε, Βεβαίω χωράνε βελτιώσεις όπως είπατε και εσείς και το, και, και, και το Κοινοβούλιο μπορεί να βοηθήσει για να συμφωνήσει καλύτερα το Συμβούλιο. Ευχαριστώ. Ε, molto brevemente, ε, Πολύ σύντομα. Στην προηγούμενη συνεδρίαση της COSAC Παρατήρησα ότι η αντιπροσωπεία των αισθανών βουλευτών, τους οποίους ε, μάλιστα είδαμε και στο Ευρωκοινοβούλιο, ήταν ιδιαίτερα δυναμική όσον αφορούσε τις υποχρεωτικές προσωστώσεις. Έλεγε ναι, είναι δίκαιο να αντιμετωπιστεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο το πρόβλημα, η διαχείριση των μεταναστευτικών ροών, αλλά μετά με βάση την αρχή της επικορικότητας θα πρέπει να σεβαστούμε την κυριαρχία των κρατών μελών, άρα εμείς αποφασίζουμε αν, πότε και, αν, και, και πόσους θα υποδεχτούμε. Κάτι που θέλω να προσθέσω ε, σε όσα είπαν ήδη οι συνάδελφοι, τα, οι ποσοστώσεις, ακόμα και αυτές οι υποχρεωτικές, δεν μ' αρέσουν και πολύ ε, για να συνεννοούμαστε. Σέβονται τις αρχές ε, της αναλογικότητας. Φυσικά ε, μετράται η δημογραφία, ο πληθυσμός, το ΑΕΠ, το εγχώριο προϊόν και οι πραγματικές δυνατότητες του κάθε κράτος μέλος να υποδεχτεί μετανάστες και μετά σε σχέση με, την, με τη δυνατότητα επιλογής. Είναι κάτι που εμείς το ζητήσαμε. Το ζητήσαμε για να αποφύγουμε τις δευτερογενείς μετακινήσεις μετά, δηλαδή εντός το ζητήσαμε μέσα στο οπτική της ε, κοινωνικής ε, ένταξης, γιατί πολύ συχνά ε, δεχόμαστε αλλά δεν εντάσσουμε στις κοινωνίες μας και έπειτα δημιουργούνται μόνιμες εντάσεις ανάμεσα στους πολίτες που υποδέχονται και αυτούς που έχουν φτάσει, καταφτάσει. Τώρα η ερώτηση των ερωτήσεων, η καταληκτική, τελευταία, εσχάτη, ποιος. Έτσι μ' αρέσετε. Λοιπόν, εσείς, παρακαλώ. Εσείς θα, θα τερματίσετε όλες τις ερωτήσεις. Η μητέρα όλων των ερωτήσεων. Η Πορτογαλίδα. Ε, ε όρους ανθρωπιστικούς. Α, Σοφία Μαρένα από την Πορτογαλία. Ε, σε όρους ανθρωπιστικούς αλλά και ασφαλείας, όπως ακούμε, δεν θα είχε περισσότερο νόημα να έχουμε κέντρα όπου συμμετέχουν τα κράτη-μέλη, Ευρωπαϊκή Επιτροπή και διάφοροι άλλοι οργανισμοί στις γειτονικές χώρες, εκεί που βρίσκονται οι περισσότεροι πρόσφυγες. Να μην περιμένουμε να φτάνουν εδώ ή να πεθαίνουν, να πνίγονται προσπαθώντας να φτάσουν στην Ευρώπη. Δεν θα σήμαινε αυτό, δεν θα έχει περισσότερο νόημα, εν πάση περιπτώσει. Αυτό που, μπορώ να, αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι πριν από έξι μήνες όταν προσωπικά έθεσα το θέμα να ιδρυθούν τα hot spots στα παράλια της Τουρκίας αντιμετωπίζοντας το μεγάλο κύμα των ε, προσφύγων. Δεν μπορούσε αυτό να υποθεί, ε, θεωρεί το ε, εκτός αντικειμένου. Τώρα πληροφορούμε ότι αδρά σιγά σιγά έχει μπει στο τραπέζι μιας κάποιας συζήτησης. Εκτιμώ ότι χρειάζεται πολλής χρόνος για γιατί αντιλαμβάνεστε ότι στα πλαίσια μιας συνενετικής πολιτικής μπορεί και διπλωματικών σχέσεων να τεθεί, δεν μπορεί συγκρουσιακά Άρα ίσως να έχει οριμάσει η ιδέα του να μπει στο τραπέζι και αυτό σαν μια ε, διαχείριση κατεύθυνσης οριστικής του προβλήματος. Ευχαριστώ. Μαλίν Διόκ. Όχι. Δεν πρέπει να έχουμε στρατόπεδα εκτός της Ένωσης που να τους ε, σταματάμε. Όχι γιατί αυτό μας λένε οι οργανισμοί ανθρωπίνων δικαιωμάτων και πρέπει να το πάρουμε σοβαρά. Γι' αυτό και οι Αφρικανοί εταίροι μας ε, το απέρριψαν. Γιατί ήταν ε, επιτάπητος ε, στη Βαλέτα και οι Αφρικανοί μας είπαν όχι δεν θα κάνουμε τη βρωμοδουλειά σας. Γιατί η πραγματικότητα είναι πως η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν τα παίρνει τόσο σοβαρά τα ανθρώπινα δικαιώματα όταν κατηγείται εκτό των σύνορων. Νομίζω λοιπόν πω θα ήταν μια επικίνδυνη εξέλιξη. Η δική μου θέση είναι διαφορετική. Πρέπει να δώσουμε τη δυνατότητα να ανοίξουν hot spot, αλλά να, και δυνατότητα να μπορούμε να υποδεχτούμε τους ανθρώπους, ε, γιατί πρόσφατα ε, ε, επισκέφθηκα διάφορες χώρες, όπως η Μπουρκίνα Φάσο, όπου επευλέψαμε τις εκλογές, έχουν γίνει διάφορα πραξικοπήματα, η κατάσταση είναι δραματική, αλλά και σε άλλα μέρη όπου, όπου προέρχονται μετανάστες. Εγώ λέω, δεν μπορούμε να κλείνουμε τα μάτια απέναντι σε κανέναν. Όταν δηλαδή ένα κράτος δεν αναλαμβάνει την ευθύνη και να πει ότι μπορώ να έχω συγκεκριμένα σημεία όπου να υποδεχτώ και να δημιουργήσουμε και ανθρωπιστικούς διαδρόμου, αλλά όχι ε, στρατόπεδα κράτηση. και σε αυτό πρέπει να προσέξουμε. Αυτό σημαίνει ότι δεν θέλει να ασχοληθεί με το θέμα. Γι' αυτό λέω, δεν μπορούμε να παραβλέπουμε το γεγονό ότι υπάρχουν άνθρωποι από την άλλη μεριά. Και αν μιλάμε για την Ευρωπαϊκή Ένωση, α μιλήσουμε και για την Αφρικανική Ένωση. Μα τι κάνει η Αφρικανική Ένωση όταν μιλάμε για ευθύνε, θα πρέπει να μιλήσουμε για συνυπευθυνότητα. Γιατί αυτή τη στιγμή το θέμα του μεταναστευτικού φαινομένου Ηνωμένων. ναι, απασχολεί την Ευρώπη και έχει ευθύνε, αλλά ε, αφορά και του θύνοντε σε άλλα μέρη, όπου ανα πάσα στιγμή θέλουν να πάρουν την εξουσία, αλλά τελικά μένουν ε, και απλά και μόνο είναι τις, ε, και να παραμείνουν ακόμα περισσότερο. Αυτό είναι ο στόχο του. Αλλάζουν το Σύνταγμα και ξανά μανά για να ξαναεκλεγούν. Αυτό που έλειψε λοιπόν στη Μάλτα είναι αυτό. Τελείωσαν τα πολλά λόγια. Τώρα πρέπει να περάσουμε στι πράξει, σε συγκεκριμένα πράγματα. Και αυτά τα συγκεκριμένα βήματα δεν τα βλέπω ούτε από την άλλη πλευρά. Πρέπει να μπορέσουμε να καλέσουμε όσους ε, ε, ε γκρινιάζουν να μας πούν γιατί αυτός ο κόσμος έβγαινε από τη χώρα σας και πρέπει όλα να τα δούμε ξανά, να ξαναδούμε τις συμφωνίες τις εμπορικές, τις οικονομικές, τα όσα αφορούν όλους τους τομείς. Γι' αυτό και λέω, ε, όταν υπάρχει κόσμος στους δρόμους, κάποιος τους έχει διώξει. Γιατί και πώς. Ναι, συγγνώμη, μπορώ να κάνω μια συμπληρωματική. Εγώ ρωτάω, γιατί να μην μπορεί κανείς να ζητήσει το άσυλο στην Τουρκία ή στο Λίβανο. Καταλαβαίνω αυτό που μου είπατε, ότι όταν γίνεται... Πρέπει κάποιος να φτάσει εδώ για να ζητήσει άσυλο, αλλά δεν υπάρχει νόμιμος δρόμος για να φτάσει. Αυτό ήταν το ερώτημα. Με αυτή την έννοια το ρώτησα. Ναι, εγώ να απαντήσω σε όσα μόλις είπατε. Ακριβώ το πρόβλημα είναι ότι δεν υπάρχουν νόμιμε εναλλακτικέ. Να μπορεί δηλαδή να έρθει κανεί νόμιμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Γι' αυτό και οι καταβλισμοί των προσφύγων είναι προσωρινέ λύσει. Δεν είναι λύσει όμως. Εμείς πρέπει να παρέχουμε μια νομική εναλλακτική που αυτή τη στιγμή λείπει. Ε, όταν αρχικά μιλούσαμε για αναθεώρηση του κανονισμού του Δουβλίνου, ο Επίτροπος Αβραμόπουλος έλεγε όχι, είναι τώρα νωρί, είναι πρωίμο, όλα μια χαρά πάνε. Όπως και διάφοροι συνάδελφοι ήταν κατά. Σήμερα όμως ε, ο ίδιος ο Γιούγκερ είπε ότι είναι απαραίτητο να ξαναδούμε το Δουβλίνο. Το είπε ο Γιούγκερ, το είπε ο Τίμερμαν, το λέει και ο Αβραμόπουλος. Για μας αυτό είναι πολύ ικανοποιητικό. Οι καταβλισμοί προσφύγων μπορούν να είναι πολύ επικίνδυνοι. Γιατί, Γιατί μπορεί να θέσουν σε κίνδυνο την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων και επειδή αν δεν γίνουν σωστή διαχείριση παρισφρίουν εγκληματικέ οργανώσεις όπως γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά. Και γι' αυτό η λύση θα έπρεπε να είναι οι νόμιμε οδοί πρόσβαση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. No, um, there is already... Κοιτάξτε, Ήδη ακούμε για αποθήσεις ε, στα hotspot που έχουν δημιουργηθεί μέσα στην Ευρώπη. Πριν φτάσουμε λοιπόν σε μια ασφαλή κατάσταση όπου θα γίνεται σεβαστό το δικαίωμα στο άσυλο, δεν νομίζω δηλαδή. Είναι αυτό που σας είπα, ο Τούσκ θέλει να, να θέσει εξωτερικά τα σύνορα. Τεχνοκρατικά θα μπορούσε να είναι λύση, αλλά στον πραγματικό κόσμο δεν νομίζω. Okay, but quick. Ε, αλλά σύντομα. Δηλαδή προτιμάτε αυτοί οι άνθρωποι να μπαίνουν στις βάρκες. Να μπαίνουν στις βάρκες, ε, να ρισκάρουν τις ζωές τους ε, και να έρθουν στην Ελλάδα και στην Ιταλία και να πληρώνουν. Αντί να μείνουν στην Τουρκία και το Λίβανο και να έρθουν από εκεί. Όχι, εμείς στην αριστερά είμαστε υπέρ νομίμων διόδων. Θέλουμε δηλαδή να υπάρχει δυνατότητα μιας βίζας για να μπαίνουν οι άνθρωποι νομίμως και να ε, εξεταστεί έτσι τους ένα κάρτος μέλος. Νομίζω ε, θα συνεχίσετε στο Κοινοβουλίο. Μια φορά δεν το κάνετε γιατί είναι σχεδόν άδειο. Σας ευχαριστώ, τελειώσαμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ σας ευχαριστώ και τους Γερμηνείς. Λοιπόν, καλώς ήρθατε στις Βρυξέλλες ε, και τα λέμε για σας.